uno vale και κύριοι, θα επιθυμούσαμε να αρχίσουμε γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο σήμερα το απόγευμα. Σα καλωσορίζω όλου θερμότατα στην ακρόαση αυτή και χαίρομαι που παρευρίσκεται ο επίτροπο Sports. Καλωσορίζω και ε, τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Κλουτσίνσκας. Ε, ε, καλωσορίζω ορίζω τους συναδέλφους και όλους τους ενδιαφερομένους που ήρθαν στην ακρόασή μας για του επίσημου ελέγχου σε ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα. Έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα ασφαλείας στην προστασία των φυτών, ζώων και ανθρώπων, αλλά θα πρέπει να λειτουργεί καλά και η αγορά. Και τα δύο είναι σημαντικά μελήματα και για να είναι εξασφαλισμένα και τα δύο, το κοινοτικό δίκαιο έχει εναρμονισμένες προδιαγραφές σε σχέση με κινδύνους που μπορούν να εμφανιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της διατροφικής αλυσίδας. Δεν είναι τόσο παλιός αυτός ο όρος διατροφική αλυσίδα και εδώ χρησιμοποιείται και με την ευρύτατη έννοια. Αυτή η αλυσίδα των τροφίμων έχει να κάνει με όλες τις μεθόδους, δραστηριότητες, προϊόντα ε, που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, διάθεση και χειρισμούς με τρόφιμα. Το 2004 μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προχώρησαν σε έγκριση ε, κανονισμού για τους ε, επισήμους ελέγχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μετά από τόσα χρόνια έχει κάνει πρόταση ε, για ανανέωση του κανονισμού, αναδιατύπωσή του μάλλον, ε, που καλείται να αντικαταστήσει και τα άλλα νομοθετήματα για να έχουμε ε, ένα διαφανές πλαίσιο αηφόρο πλέον θεσμικό και που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Είναι σημαντικό αυτό κυρίως για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της Ένωσης. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τμήμα μιας δέσμης μέτρων ε, που τώρα το κεκτημένο καλείται να ε, εξυγχρονιστεί και για την προστασία των ζώων και των φυτών και ε, του πολλαπλασιαστικού λεγόμενου υλικού. Χαίρομαι που βλέπω εδώ εκπροσώπους της διοίκησης, της πράξης αλλά και των καταναλωτών. Ε, θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στο Μάριο Πεδίο, τον εισηγητή μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος επί της ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος για να αφήσω χώρο και χρόνο στη συζήτηση και τις παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές και τους ε, συμμετέχοντες για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα των επισήμων ελέγχων που εντάσσεται σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και αφορά ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Λιθουανική Προεδρία, τον Επίτροπο Πόργ για τον επικοδομητικό διάλογο που προωθείται μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, πολυσχηδούς νομοθετικής πρότασης. Πρόκειται για πληθώρα τομέων και δεν θα μας απασχολήσουν όλοι στη σημερινή συνάντηση, όχι γιατί είναι ίσονος σημασίας, αλλά για λόγους καθαρά έλλειψης χρόνου. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο τομέας της διατροφικής αλυσίδας είναι ύψης της σημασίας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απασχολεί 48 εκατομμύρια εργαζομένους με ένα ε, τζίρο 150 δις Τα παράγωγα προϊόντα Ε, χαίρουν υψηλού ε, επίπεδου ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια ενός ειδικού νομοθετικού πλαισίου. Παρ' όλα αυτά, μας έπληξαν πολλά σκάνδαλα κατά τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως ε, και το κρέας αλόγου ήταν το τελευταίο από αυτά τα σκάνδαλα που γνωρίζετε. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο ελέγχων και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ για αυτή την εργασία που δεν ήταν καθόλου εύκολη τα τελευταία χρόνια για να φτάσουμε σε μια νέα πρόταση. Ο κανονισμός 882 του 2004 αφήνει περιθώρια ερμηνείας από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει εν ώψη του μελλοντικού κανονισμού να διασαφίσουμε το περιεχόμενο αυτού του κανονιστικού πλαισίου. Οπωσδήποτε η κατεξιοδότηση πράξης μπορούν να αποδυναμώσουν το κείμενο, αλλά εδώ θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Στόχος είναι να ακούσουμε και είμαι τους εμπειρογνώμονες και είμαι πεπισμένος ότι οι συζητήσεις και οι παρουσιάσεις με την εκπροσώπηση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ενώσεων και φορέων θα μας βοηθήσουν για να δούμε την οπτική εκείνων που σχετίζονται, που ασχολούνται μάλλον με την εφαρμογή αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Να γνωρίσουμε τις απόψεις τους έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ε, υπερβούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριο Πυρίλου. Ε, η Ράιμερ, συγγνώμη, έχει το λόγο εξ ονόματος της ε, Επιτροπής Γεωργίας που γνωμοδοτεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που ασχολούμαστε ε, με αυτούς τους επισήμους ελέγχους ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και θέλουμε να ε, ομοιογενοποιήσουμε, να ενιοποιήσουμε και να απλουστεύσουμε και να εξυγχρονίσουμε αυτό το σύστημα. Τα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, τα διάφορα προβλήματα, γι' αυτό η δραστηριότητα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ θα πρέπει να χαιρετιστεί και να καλωσοριστεί. Θα πρέπει να προσέξουμε το εξής, να τηρούμε ε, το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για τα τρόφιμα, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να τη διατηρήσουμε στη συνέχεια και δεν θα πρέπει να λησπονούμε ότι πρέπει να στραφούμε και προς τα έξω και να ε, εξασφαλίζουμε και την εμπιστοσύνη των τρίτων κρατών ε, τους επίσημους ελέγχους μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Θα πρέπει να παραμένει η ασφάλεια τρομή εγγυημένη, το κράτος βεβαίως να εγγυάται αυτή την ποιότητα. Τι εννοώ. Βεβαίως θα πρέπει οι επιχειρήσεις και οι εταιρείε να συμμετέχουν στον έλεγχο των τροφίμων, αλλά δεν θα πρέπει να την επιβαρύνουμε ιδιαιτέρως, ούτε θα πρέπει αυτή η κρατική αρμοδιότητα να υποκατασταθεί από μια ιδιωτική. Ε, να εξευρεθεί εκεί κάποια ισορροπία. Χαίρομαι για τη σημερινή ακρόαση. Θα ακούσουμε διάφορους εμπειρογνώμονες και ειδικού ε, για να μας πούν τι μπορούμε να βελτιώσουμε στα κείμενα ε, που ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία έτσι ώστε να είναι κάπως ικανοποιημένες όλες οι πλευρές και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια όπως είπαμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, και τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία και ε, χαίρομαι για τη συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια και εύχομαι καλή επιτυχία στην ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ράιμερς και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεβίντα Κιλουτσίνσκα, που είναι αναπληρωτή πρόεδρο τη Αρμόδιας ομάδα εργασία του Συμβουλίου Ψήμων Ελέγχων και εκπρόσωπο τη Λιθουανικής Προεδρία. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Ισηγητά, Περίλο, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, καταρχήν εξ ονόματος ε, του κυρίου Γιούκνα, του Υπουργού Γεωργίας από τη Λιθουανία, θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω και να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του. Όπως ξέρετε, η Λιθουανία αντιμετωπίζει προβλήματα με τη Ρωσία εξαιτίας της απαγόρευσης των ε, γαλακτοκομικών προϊόντων και δυστυχώς ο Υπουργός μας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω σήμερα για να επιβεβαιώσω τη σημασία που προσδίδουμε σε αυτό το θέμα και το μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησης της εργασίας σας έτσι θα μπορέσουμε να ακούσουμε τα πρωταρχικά προκαταρκτικά σχόλια των κρατών μελών και παράλληλα μας ενδιαφέρει η άποψη των εμπλεκομένων φορέων, εκείνων δηλαδή που συνεργάστηκαν με την Κόπα Κοτζέκα μαζί με την Ιρλανδική Προεδρία τον Μάιο, πέρσι το Μάιο και έτσι εξέτασαν τις λεπτομέρειες της πρότασης. Η πρόταση αυτή είναι μέρος του πακέτου μέσα στα πλαίσια του αναπαραγωγικού υλικού, ε, υγείας των ζώων και ποιότητας των ζωοτροφών, καθώς και δαπανών στον τομέα αυτό που παρουσιάστηκε πέρσι το Μάιο. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, σωστή παρουσίαση της νομοθεσίας, τη βασική δηλαδή νομοθεσία που θα πρέπει να ισχύσει σε αυτό το τομέα, ιδιαίτερα για τα τρόφιμα και τις τροφές, για την, ε, το αναπαρογικό υλικό, την ε, ζωική ευεξία και την υγεία και υγιεινή όσον αφορά τα ζώα και τα φύτα. Η Λιθουανική Προεδρία θα ήθελε να επιτελέσει μεγάλη πρόοδο στο Συμβούλιο, σε αυτό το τομέα, εργαστήκαμε πολύ σκληρά για... στον τομέα των ταπανών, κείμενο το οποίο θα εγκριθεί τάχιστα ως προς τις, ε, επίση, τους επίσημους ελέγχους και τις τεχνικές προδιαγραφές και ελέγχους. Πρόκειται για μία τρέχουσα διαδικασία και η Προεδρία θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για να μπορέσουν να γίνουν οι συζητήσεις όπως πρέπει. Ως ε, μέρος του πακέτου και επειδή πρόκειται για ένα πακέτο θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνεκτικότητα και να γίνουν και εσωτερικές διαβουλεύσεις και συντονισμός με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα έχουμε μια εντολή μέχρι το τέλος του έτους, όμως θα γίνουν ε, τεχνικές ε, ε, διερευνήσεις για να προωθήσουμε την εργασία του Συμβουλίου. Βεβαίως, ως Προεδρία θα είμαστε σε επαφή μαζί σας, κύριε Πυρίλο, για να σας μιλήσουμε για την πρόοδο των εργασιών στο Συμβουλίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλουτσίνσκαν, πολύ καλή παρουσίαση και πολύ ουσιαστική. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπό μας, τον κύριο Μπόρτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να προσπαθήσω να εξηγήσω αυτή την ευρύτατη νομοθεσία. Δεν πρόκειται για ένα απλό νομοθέτημα, πρόκειται για ένα πακέτο το οποίο συμπεριλαμβάνει την υγεία των ε, ζώων, την φυτική υγεία, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, τους επίσημους ελέγχους και βεβαίως τη διαχείριση των δαπανών της ε, Κομισιόν στους τομείς αυτούς. Περιτώ να πω ότι η επίσημη έλεγχη είναι ουσιαστική εκ των όνου κάνε, αν θέλουμε να κρατήσουμε ακέραιη τη φήμη μας ως μια περιοχή του κόσμου που έχει τις πιο, τους πιο αυστηρούς κανόνες για την ε, διατροφική αλυσίδα παρά τα γεγονότα, τα σκάνδαλα που ε, από καιρούς καιρό ξεσπάνε. Αυτοί οι κανόνες υπάρχουν, ε, εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη σε όλους τους τομείς της γεωργοδιατροφικής αλυσίδας με υγιή, δίκαιο και ανεξάρτητο τρόπο και αυτό είναι σημαντικό αυτοί οι έλεγχοι από τα κράτη-μέλη να συμπληρώνονται από κατάλληλους ελέγχους, από εμπειρογνώμονες της Κομισιόν ε, που ελέγχουν τους εθνικούς ε, ελέγχους. Αυτό το πακέτο ξεκίνησε, δρομολογήθηκε όπως τα ξέρετε στις 6 Μαΐου, φαντάζομαι ότι όλοι θα είστε εξοικειωμένοι με το περιεχόμενό του και Ο κύριος Πυρίλα ανέφερε κάποια πράγματα και θέλω να σας πω ότι το πακέτο τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τις αντιδράσεις που έγιναν σε σχέση με κάποια σκάνδαλα που δεν ήταν σοβαρά πράγματα, επρόκειτο για κάποιες απάτες στην πραγματικότητα. Προτείνουμε λοιπόν για πρώτη φορά σε αυτήν την νομοθεσία τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις όταν συμβούν στο μέλλον ε, κάποια προβλήματα οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που να αντικατοπτρίζουν τα παράνομα κέρδη που έχουν δρέψει αυτοί οι εμπορευόμενοι οι οποίοι αποφάσισαν να αγνοήσουν τον νόμο, να παραβιάσουν τον νόμο. Όταν υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με έλεγχο του DNA σε όλα τα κράτη-μέλη για να δούμε κατά πόσο υπάρχει αλογίσιο κρέας στο βόλιο ή κατά πόσον υπάρχουν ε, αντιφλεγμονώδη φάρμακα ε, στο κρέας που δεν θα έπρεπε να έχει μπει στη διατροφική αλυσίδα. Αυτό θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Όταν κάναμε αυτούς τους ελέγχους ε, DNA με βάση τις συστάσεις, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη υπερέβησαν το στόχο που είχαμε ε, συστήσεις ό,τι αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων, τον αριθμό των ελέγχων. Οι μεγάλες χώρες, ας πούμε, ε, σε αυτές είχαμε συστήσει να κάνουν 250 τεστ και έκαναν 800 ε, δοκιμές, 250, 800 δοκιμές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, όλα τα άλογα ελέγχθηκαν και όχι μόνο κάποια. Οι αντιδράσει λοιπόν ήταν πολύ θετικές και τώρα προσπαθούμε να έχουμε ένα νομικό περίβλημα σε αυτές τις δράσεις που ούτως ή άλλως προωθούν τα κράτη-μέλη, κομισιόν κτλ. μετά από το σκάνδαλο με το κρέας του αλογίσιο. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα να διευκρινίσω γιατί φαντάζομαι ότι θα προκαλέσουν συζητήσεις στο Κοινοβούλιο αλλά και εκτός του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο θέματα από αυτή την νομοθεσία, τη χρηματοδότηση και το σύνηθες επίμαχο θέμα των καταξιοδότηση πράξεων. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων, θα ήθελα να σας πω ότι η βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συστήματος και των εθνικών ελεγκτικών ε, υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες να τους διενεργήσουν είναι το διακύβευμα εδώ και δεν μπορούμε να υποσκάψουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών για να κάνουν ε, αποτελεσματικούς ελέγχους, ε, γιατί αυτό θα μας ε, άφηνε εκτεθειμένους σε κινδύνους για σοβαρούς, σοβαρά σκάνδαλα στον τομέα των τροφίμων. Ε, υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια τα οποία ε, λόγω της οικονομικής κρίσης οδηγούν σε μείωση στο επίπεδο των ελέγχων ε, σε κάποια, αν όχι σε όλα τα, στα περισσότερα κράτη-μέλη. Και φυσικά αυτό δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών και για την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού συστήματος συνολικά. Λοιπόν, για τα τέλη που ε, εφαρμόζονται τώρα στους ελέγχους. Θα τα εφαρμόσουμε τώρα με αυτή την νομοθεσία στους περισσότερους τομείς ε, της ε, γεωργοδιατροφικής αλυσίδας. Και με βάση το σχέδιο των κανόνων ε, θεωρούμε ε, ότι όλη η αλυσίδα των επίσημων ελέγχων αποτελεί μια πολύτιμη υπηρεσία με προσθέμενη αξία. Ξέρω ότι κάποιοι ανησυχούν ότι αυτή η κίνηση θα δημιουργήσει αύξηση του κόστους και δεν θα δώσει κίνητρα στις υπηρεσίες επιθεωρήσεων και ελέγχων για να κάνουν ε, επίσημους ελέγχους. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η αλλαγή δεν προτείνεται μεμονωμένα και δεν θα πρέπει να εξεταστεί απομονωμένα. Γιατί αυτό που προτείνει η Κομισιόν σε αυτό το πακέτο σε ό,τι αφορά τους επίσημους ελέγχους και τα τέλη είναι να υπάρχουν ε, πιο αυστηρές προϋποθέσεις ε, διαφάνειας, λογοδοσίας, από τις ε, ελεκτικές αρχές τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για το πώς ε, χρηματοδοτούνται οι έλεγχοι, για το πώς ε, υπολογίζονται τα τέλη, πώς δαπανώνται αυτά τα ποσά και για κάποιες διαθετήσεις για να αποφύγουμε την αναποτελεσματική χρήση των πόρων που συλλέγονται μέσω των τελών. Επομένως, θα διευρύνουμε τη συλλογή των υποχρεωτικών τελών για σε βασικές δραστηριότητες του γεωργοδιατροφικού τομέα και με αυτό θα εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του επίσημου συστήματος ελέγχων, ε, απομονώνοντάς τον από τις ε, τοπικές ε, δημοσιονομικές αποφάσεις, αυξάνοντας παράλληλα με την αύξηση της, ε, των υποχρεωτικών τελών, με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε την, τη λογοδοσία των ε, αρχών που διεργούν τους ελέγχους για το πώς προβαίνουν σε αυτούς τους ελέγχους. Όλες οι μικρές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς ε, του κλάδου ε, εξαιρούνται όμως από την υποχρέωση να καταβάλουν τέλη και αυτό συνάδει με την πολιτική της Κομισιόν να μειώσει το βάρος και να προσαρμόσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στις ανάγκες των μικροεπιχειρήσεων. Κατεξοδότηση πράξης. Ξέρω ότι η Κομισιόν όταν προτείνει ένα νομοθετικό πακέτο, προτείνει, ε, και όταν μάλιστα αυτό αφορά πέντε ή έξι τομείς, πάντα υπάρχουν α, ε, κατεξοδότηση πράξη. Ξέρετε τι αλλεργίες αυτές, όπως και τα εθνικά κοινοβούλια. Κάθε φορά που το κοινοβούλιο ε, χωρεί αρμοδιότητες στην ε, κυβέρνηση, στην εκτελεστική εξουσία, ε, αυτό συνοδεύεται με μια σειρά από προθέσει. Όταν ήμουν φοιτητή νομική θυμάμαι, ο Τζουλ, ένα αγγλικό βιβλίο συνταγματικού δικαίου έλεγε ότι οι κανονισμοί βάζουν σάρκα στην ξεραήλα των οστών του νόμου. Οποιαδήποτε νομοθεσία χρειάζεται κατεξουσιοδότηση νομοθετήματα, ούτω ώστε να συμπληρωθούν τα κενά, ούτω ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία, ούτω ώστε να μην βαρύνουμε το κύριο σώμα της του νομοθετήματος με περιττές λεπτομέρειες. Φανταστείτε λοιπόν, αν δεν, αν δεν υπήρχε δευτερογενή νομοθεσία, αν υπήρχαν κατεξουσιοδότηση πράξης, θα έπρεπε όλα τα στοιχεία, όλες τις λεπτομέρειες να τις βάλουμε στο διατακτικό και να το βαρύνουμε θα ήταν απίστευτα σχολαστικό αυτό το κείμενο και επίσης δεν θα μας εξασφάλιζε την απαραίτητη ευελιξία, ούτω ώστε να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις ε, και ξέρουμε πολύ καλά ούτως ή άλλως ότι σε ό,τι αφορά την, ε, της πράξη υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος από το Συμβούλιο. Αν επομένως προκύψουν νέοι κίνδυνοι ή οποιοδήποτε πρόβλημα, θα υπάρχει μέσω της νομοθεσίας αυτής, μέσω των κατευθυντών της υπράξεων, θα μπορούμε να απαντήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιους κινδύνους. Φυσικά όμως το μπαλάκι είναι στα χέρια, είναι στο γήπεδο των συνομοθετών σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Σας κάνω έκκληση όμως, αν θέλετε να αυξήσετε τις προϋποθέσεις ε, για τις ε, κατευθυντικές πράξεις να το κάνετε, αλλά αν τις καταργήσετε γιατί για τέτοια ε, λεπτά θέματα είναι εκ των όνου κάνευ. Αλλά αυτό είναι μία σύσταση της Κομισιόν. Επομένως, να πω και κάποια άλλα από τα ωφέλη με τη νέα νομοθεσία. Καταρχάς, έλεγχη στα σύνορα. Έχω ακούσει παράπονο ότι μερικές φορές είμαστε πιο αυστηροί με τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είμαστε τόσο αυστηροί με παραγωγούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξάγουν το προϊόν τους στην Ευρώπη, σε εμά. Με αυτή την νομοθεσία νομίζω, νομίζω ότι θα έχουμε ε, μια πιο αποτελεσματική κατανομή του βάρους ε, των ελέγχων και αυτό θα είναι καλό και για τους εισαγωγείς, για τους παραγωγούς κτλ. Οι εισαγωγείς λοιπόν θα υποφεληθούν από απλούστερη ε, από ένα απλούστερο ε, μηχανισμό ε, για τους ελέγχους στα σύνορα. Απλούστερες διαδικασίες, ε, ένα ενιαίο έγγραφο για τα, για τα ένα ενιαίο έντυπο για τα έγγραφα και ηλεκτρονικά έγγραφα, έντυπα γενικά. Το νέο σύστημα θα εξασφαλίσει ότι οι διαθετήσεις αυτές στα σύνορά μας προσαρμόζονται στο επίπεδο του κινδύνου ε, που συνδέονται με τα τρόφιμα αυτά που προέρχονται από τις τρίτες χώρες. Λοιπόν, οι καταναλωτές επίσης και οι τίμοι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι το τμήμα της προσπάθειας του ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές θα πηγαίνουν σε συγκεκριμένες προσπάθειες ελέγχου για να εντοπίσουν τις αποπρόθεση παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων και τις παραπλανητικές πρακτικές, με άλλα λόγια την απάτη. Ε, το πρόσφατο σκάνδαλο με το λογίσιο κρέας ε, έδειξε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή σε οποιαδήποτε σημάδια, μηνύματα έχουμε για παράνομες πρακτικές παρά να αντιδρούμε εκ των, υστέρων. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζουμε και θα καταργούμε, θα ακυρώνουμε οποιαδήποτε τέτοια άτιμη συμπεριφορά το συντομότερο δυνατό. Οι νέοι κανόνες επίσης θα επιβάλλουν και οικονομικές κυρώσεις. Και βεβαίω, όσοι κάνουν τέτοιε απάτες τα πληρώνουν. Επίσης, ε, τα βελτιωμένα αυτά εργαλεία για, τους, ε, τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών θα μας βοηθήσουν ε, ούτω ώστε οι απάτε και η μη συμμόρφωση που επηρεάζουν πολλά κράτη-μέλη να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Πιστεύω, πιστεύω ότι αυτά τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν με αυτήν την νομοθεσία στο μέλλον Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και σας υπενθυμίζω ότι οι υπηρεσίες μου είναι στην απόλυτη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Το θέμα αυτό ε, δημιουργεί πολλά πάθη η διατροφική ασφάλεια, η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μας ενδιαφέρει είναι τα σκάνδαλα αυτά. Να μην έχουμε πλέον άλλα σκάνδαλα που ε, να ανακύψουν στον τομέα του κρέατος επειδή δεν εφαρμόστηκε το νομοθετικό πλαίσιο. Το ζήτημα είναι κατά πόσο έχουμε φτάσει στη σωστή, ε, σε μια ισορροπία ως προς τον νόμο και την εφαρμογή του. Όταν μιλάμε για κατεξιοδότηση πράξης, είμαστε όλοι πολύ ευαίσθητοι, ως... υπάρχει μια ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει να υπάρχει πολιτικό input στον κανονισμό και η Κομισιόν θα πρέπει να βασιστεί σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει πολιτική συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα αυτά βρίσκονται επιτάπητος. Το θέμα αυτό είναι ευρύ και χαίρομαι που έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες σήμερα το απόγευμα για να μας εκθέσουν την άποψή του. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Horst Σνέλχαρτ, ο οποίος θα αναλάβει τον πρώτο γύρο εμπειρογνωμών, παρουσίασης των εμπειρογνωμόνων. Έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την ακρόαση και είμαι ε, ευγνώμων γιατί ο Επίτροπος είναι εδώ μαζί μας. Πριν μιλήσω επί της ουσίας, θα ήθελα να σχολιάσω τις κατεξιοδότηση πράξης. Η Επιτροπή κατέστησε απόλυτα σαφές το πλαίσιο λειτουργίας και νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε ότι δεν πρέπει να περικοπούν οι κατεξιοδότηση πράξεις και αυτό αφορά την διατύπωση, της επιμέρους διατυπώσεις τη διατύπωση ειδικά στις κατεξουδότηση πράξεις έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφισημία. Αυτό είναι το ζητούμενο για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για κατεξουδότηση πράξης και να μην επιδέχονται ερμηνείας. Κυρίες και κύριοι, το μέλλον των επίσημων ελέγχων είναι ένα ευρύ θέμα Έχουμε αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύσει αυτό το τομέα και να αναθεωρήσει τον κανονισμό 882. Αυτό ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και περιμέναμε πολύ λιγότερα. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες ε, ε, επέκτασης του νομοθετικού πλαισίου. Έχουμε πολλούς ομιλητές στο πρώτο αυτό πάνελ. Ο Έρικ Πουντελέ είναι εδώ μαζί μας που είναι ο Διευθυντής ε, για την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας από την ε, Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, ο Μάικλ Σκάνελ που είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, κάθεται δίπλα του, ο δόκτωρ Μάρτιν Χάρτμαν που ήταν πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου ε, επισήμων κτηνιάτρων και αυτός κάθεται στην πρώτη σειρά. Ο δόκτωρ Σίλβιο Μπορέλο Νομίζω ότι κάθεστε σωστά και με τη σωστή σειρά και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ο δόκτωρ Σίλβιο Μπορέλο είναι Γενικός Διευθυντής από το Υπουργείο Υγείας, την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Ιταλίας. Έχουμε και από το Ηνωμένο Βασίλειο διάφορες μελέτες. Ε, δεν έχουν έρθει όλοι όμως. Ε, ο Διευθυντής ε, από τη Γενική Διεύθυνση Διατροφής στο Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Δεν έχει έρθει ακόμα κύριος Λοϊκεβά και παραμονές ε, των, της ακρόασης ε, είχαμε και επαφές με συναδέλφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και δυστυχώς λόγω του λουκέτου στην Αμερικανική κυβέρνηση δεν μπόρεσε να έρθει κανένας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε, οι περικοπέ πρέπει να γίνονται γέρο και ε, όχι κατόπιν εορτή, γιατί δεν μπορούν να έρθουν εμπειρογνώμονε στην Ευρώπη εκτό όλων των άλλων. Επίση, η αρμόδια ε, καναδική αρχή ε, έχει προετοιμάσει ε, την παρουσίαση σε βίντεο και powerpoint τα έχετε λάβει την περασμένη εβδομάδα και έχει καταφέρει να έρθει η κυρία που εκπροσωπεί τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σας καλωσορίζω και χαίρομαι που ήρθατε. Θα είναι η συζήτηση φαντάζομαι ε, αρκετά ανοιχτή και ειλικρινής. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τους εμπειρογνώμονες να λάβουν τη σειρά με, ε, τη, με το λόγο συγγνώμη, με τη σειρά που σας ανέφερα. Πρώτος ο κύριος Ερικ Πουντλέ. Ευχαριστώ. Ε, δυστυχώς είναι άχαρο το έργο μου, δηλαδή θα πρέπει επί PowerPoint να σας επαναλάβω αυτά που είπε ο Τίτροπος Πόρκ. Αλλά υπάρχει... το έγγραφο που σας έδωσα υπάρχει ένα PowerPoint. Θα παρουσιάσω κάποιες ε, διαφάνειες ε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Με αυτό το νέο κανονισμό ε, επαναλαμβάνουμε, ε, χρησιμοποιούμε τον κανονισμό του 2004, νέα χρόνια μετά, εννέα χρόνια μετά, ε, θεωρήσαμε απαραίτητο να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό του 2004, μετά από τους ελέγχους που έκαναν οι επιθεωρητές και ο Μάικλ Σκάνε θα σας μιλήσει σε λίγο στον αδελφός μου γι' αυτό, ε, αλλά και μετά από τις διάφορες κρίσεις που είχαμε μέσα αυτά τα εννέα χρόνια. Η κρίση του αλογίσιου κρέατος είναι αρκετά πρόσφατη, αλλά είχαμε και την κρίση στη Γερμανία του Εσερίχια Κόλλη ε, με 55 ασθενείς οι οποίοι κατέληξαν σε ανάλυση. αιμοκάθαρση. Ε, αυτή η κρίση του 2002 ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να συντάξουμε αυτόν τον κανονισμό. Αυτό οφειλόταν σε ε, έλλειψη ελέγχων στις ε, εισαγωγές και στην έλλειψη επιτόπιων ελέγχων. Ήταν μια μικροεπιχείρηση. Καμιά το δεκαριά άτομα πολύ σε αυτή η γερμανική επιχείρηση η αιστεία ας πούμε, του, της αρρώστιας ε, προέρχονταν από αυτή την ε, εταιρεία. Και αυτό μπορεί να έχει πολύ σημαντικές ε, επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία βέβαια. Ο στόχος του νέου κανονισμού είναι να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή του προηγούμενου κανονισμού του 2004 σε όλη την γεωργοδιατροφική αλυσίδα, γιατί υπήρχαν τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονταν από τον παλιό κανονισμό του 2004, όπως η φυτική υγεία, οι σπόροι, ε, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, τα φυτοφάρμακα κτλ. Και θέλαμε να έχουμε κάποιους, κάποιες αρχές για τους ελέγχους σε όλους τους τομείς με τον νέο κανονισμό. Και να βάλουμε κάτι που δεν υπήρχε στον προηγούμενο κανονισμό, ένα στοιχείο το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, που είναι αυτό των μη προαναγγελθέντων ελέγχων των ευνίδιων ελέγχων. Γιατί κανονικά οι έλεγχοι θα πρέπει να αναγγέλλονται ούτω ώστε οι ε, επιχειρήσεις να ετοιμάζονται και να μπορέσουν να δεχτούν τους επιθεωρητές. Αλλά θέλουμε να κάνουμε και τέτοιους ευνίδιου ελέγχους ε, χωρίς να τους προαναγγέλουμε ε, για να αποφεύγουμε απάτες και παραβιάσεις. Επίσης, θέλαμε τους πιο ευέλικτους κανόνες, να τους συνδυάσουμε με πιο συντονισμένες δράσεις. Στο παρελθόν, μερικές φορές είχαμε συχνότητες ελέγχων που προκαθορίζονταν για κάποια είδη προϊόντων ε, και ήταν αρκετά άκαμπτο το σύστημα. Τώρα προτείνουμε όχι υποχρεωτική συχνότητα, αλλά μια ελάχιστη συχνότητα, υποχρεωτική ελάχιστη συχνότητα ελέγχων, ε, που θα καθοριστεί, ανά περίπτωση φυσικά, και με υποχρεωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ένα σημαντικό στοιχείο που δεν υπήρχε στον παλιό κανονισμό είναι να μπορούμε να οργανώνουμε σε κοινοτικό επίπεδο συντονισμένα υποχρεωτικά σχέδια. Ο Επίτροπος Μπορτ μίλησε για το συντονισμένο σχέδιο για τις για τα τεστ DNA στο βόλιο κρέας για να δούμε αν υπάρχει εκεί μέσα κρέας αλόγου. Όλα τα κράτη-μέλη, εμείς συστήσαμε στα κράτη-μέλη να κάνουν δοκιμές, να κάνουν τεστ και όλα τα κράτη-μέλη έκαναν περισσότερα τεστ. Ήταν μια σύσταση όμως. Αν ένα κράτος μέλος είχε αρνηθεί, δεν είχαμε νομικά μέσα για να το επιβάλλουμε να κάνει αυτούς τους ελέγχους, να κάνει αυτά τα τεστ. Ενώ τώρα με, το νέο, με αυτή τη νέα νομοθεσία Προβλέπουμε υποχρεωτικά σχέδια ελέγχων. Επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε την συνεργασία διοικητικής φύσεως για την εφαρμογή της νομοθεσίας μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή είναι μια από τις ομορφιές του κανονισμού αυτού. Από τα καλά στοιχεία του κανονισμού αυτού. Γιατί σήμερα όλα τα προβλήματα δεν περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος λόγω της παγκοσμιοποίησης, λόγω της ευκολίας με την οποία κυκλοφορούν τα αγαθά και της παγκοσμιοποίησης του επορίου. Πολλά κράτη-μέλη καμιά φορά εμπλέκονται ε, σε μια κρίση, ένα σκάνδαλο, ένα πρόβλημα. Και αυτό το μηχανισμό βοήθειας και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θελήσαμε να τον ενισχύσουμε τόσο ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίε, να γίνονται όλα αυτά πολύ πιο γρήγορα, γιατί δυστυχώ βλέπουμε ότι συχνά η συνεργασία σταματά στα σύνορα μεταξύ δύο κρατών μελών. Ε, και αυτό μέσα στη μεγάλη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά προφανώς δεν είναι κάτι θετικό. Ακριβώς γι' αυτό θέλησαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης, ολοκληρωμένης ενημέρωσης, που ε, υπενθυμίσει το ΡΑΣ, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, που είναι ένας μηχανισμός που ισχύει περίπου 35 χρόνια και που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ενημερώνουν μέσω της Κομισιόν όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για την παρουσία προϊόντων τα οποία δεν συμμορφούνται με τους κανόνες διατροφικής ασφάλειας. Αυτό το νέο ε, σύστημα πληροφορικής το αφιερώνουμε πιο συγκεκριμένα, δημιουργείται πιο συγκεκριμένα για τις ε, απάτες στα τρόφιμα. Επίσης, προβλέπουμε οικονομικές κυρώσεις που θα αποφασίσουν οι διοικητικοί μηχανισμοί ή οι δικαστές, πολύ πιο αποτρεπτικοί, το είπε και ο Επίτροπος, είναι πολύ λεπτό αυτό το θέμα όμως, γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να εναρμονίσει τα, τις κυρώσεις ε, που επιβάλλουν οι δικαστές όταν υπάρχει δηλαδή μία περίπτωση που εκδικάζεται σε δικαστήριο. Θέλουμε όμως αυτές οι κυρώσεις να είναι αποτρεπτικές και τουλάχιστον ανάλογες με το κέρδος που δρέπουν τα άτομα αυτά που διενεργούν αυτές τις απάτες. Κάτι άλλο, ένα άλλο διαμάντι αυτού του κανονισμού είναι ότι έχουμε ένα σύστημα ολοκληρωμένων ενσωματωμένων ελέγχων ε, στο σύνορα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες. Σήμερα για τα ζώντα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, δηλαδή ψάρι, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, έχουμε ένα τέτοιο σύστημα, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να οργανώσουν τους ελέγχους στα σύνορα για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης οποροκυπευτικά φρούτα λαχανικά ή για τα βιομηχανικά προϊόντα ζάχαρη, φερρυπίν. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εναρμονισμένο που να βασίζεται στον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει κάθε προϊόν. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων θα μας προσδιορίσει αυτόν τον κίνδυνο ανάλογα με το προϊόν και θα ενσωματώσουμε και μία διάσταση που αφορά την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στην χώρα προέλευσης. Υπάρχει και αυτό, αυτή η παράμετρος δηλαδή στο μηχανισμό. Αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχουν προϊόντα όπου θα υπάρχουν ελάχιστοι έλεγχοι κατά την εισαγωγή και θα υπάρχουν προϊόντα βεβαίως τα οποία θα ελέγχονται πολύ περισσότερο κατά την εισαγωγή. Αυτό θα υπολογίζεται ε, δυνάμει του κινδύνου, παραδείγματο χάρη τα υπολείμματα ορμονών, ε, φυτοφάρμακα, αρρώστιες μπορεί να διαβιβαστούν, να μεταδοθούν από φυτά ή προϊόντα και βεβαίως την εμπιστοσύνη που έχουμε στα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι τρίτες χώρες. Φυσικά, αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να χρηματοδοτούνται και ξέρουμε ότι οι εθνικές αρχές μειώνουν το προσωπικό τους λόγω των δυσκολιών και της ε, οικονομικής κρίσης που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, υπάρχουν μειώσεις λοιπόν σημαντικές στο προσωπικό, για να πω δραστικές σε ορισμένα που επιβάλλουν οι δημοσιονομικοί κανόνες και θεώρησαμε χρήσιμο να προτείνουμε ένα σύστημα όπου αυτοί οι έλεγχοι θα χρηματοδοτούνται από τη, τους κλάδους που υφίστανται αυτούς τους ελέγχους. Δηλαδή, όπως όλα τα κτίρια, ε, οι πολυκατοικίες που έχουν ε, ασανσέρ πληρώνουν κάποιες εταιρείες για να ελέγχουν την ασφάλεια των ε, ασανσέρ αυτών. Ένα σύστημα, λοιπόν, έχουμε προβλέψει ένα σύστημα υποχρεωτικών τελών που καλύπτει όλο το κόστος του έλεγχου που συνδέεται με το προσωπικό, με την κατάρτιση του προσωπικού, με το εργαστήριο που κάνει τους ελέγχους, με μία όμως ε, εξαίρεση για τις μικροεπιχειρήσεις. Δηλαδή αυτές που έχουν λιγότερα από 10 άτομα. Ο, Επίτροπες, ο Επίτροπος μίλησε για αυτά. Θα περάσω τώρα στη τελευταία διαφάνεια, όπου θα θέλαμε αυτή η επίσημη έλεγχη να γίνονται από κάθε κράτος μέλος μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτα διαφανές, ούτω ώστε οι διάφοροι εμπλεκόμενοι, ο κλάδος, ο γεωργοδιατροφικός, οι γεωργοί, αλλά και οι καταναλωτές να μπορούν να βλέπουν ε, προς τα που κινούνται αυτοί οι έλεγχοι, ποιο σκοπό έχουν. Και φυσικά θα υπάρχουν ε, εκθέσεις για την συμμόρφωση και μη συμμόρφωση, Και τώρα φτάνω στο συμπέρασμά μου. Σε αυτό το σχέδιο προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε μία ισορροπία ανάμεσα στους τρεις βασικούς ε, ε, στις συνιστώσεις. τους επιθεωρητές, την βιομηχανία, τον κλάδο δηλαδή, τους γεωργούς, από τους γεωργούς μέχρι τα σούπερ μάρκετ και τα εστιατόρια και η τρίτη διάσταση και πιο σημαντικοί για, την, για τους οποίους και δουλεύουμε εμείς, οι καταναλωτές. Αυτά για το νέο κείμενο, κυρία Πρόεδρε, για τους ελέγχους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή, δόκτωρα Ποντλέ. Είπατε τα βασικότερα και σίγουρα θα συζητήσουμε. Ε, είναι πολλά τα σχόλια ε, που ήδη έχω σημειώσει κι εγώ. Θα ακούσουμε πρώτο τον κύριο Σκανέλ από το Γραφείο Τροφίμων και Εκτινιατρικών Θεμάτων ε, να μας μιλήσει για την περιγραφή των πορισμάτων από αποστολές ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη-μέλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, ε, γίνονται, ε, διενεργούνται πολλά, πολλοί έλεγχοι κάθε χρόνο στα κράτη-μέλη. Δεν θα σας δώσω ε, όλα τα στοιχεία, θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία μίζων σημασίας που έχουν σημασία για τους δικούς σας ελέγχους. Και θα ήθελα να τονίσω τα ευρήματα στα διάφορα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα θέματα μπορεί να μην ανοιχνευτούν για μεγάλο ε, χρονικό διάστημα. Γι' αυτό πολλές φορές ε, δεν βλέπουμε τις ε, αδυναμίες των συστημάτων. Θα σας μιλήσω για ειδικά προβλήματα. Ένα θέμα που απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη και τις αρχές είναι το θέμα των πόρων. Αντιμετωπίζουν μεγάλα μεγάλα και πολλά αιτήματα και γι' αυτό πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα δύσκολο ζήτημα. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο με βάση τις ε, νυν οικονομικές συνιστώσεις. Θα πρέπει να γίνουν εξοικονομήσεις ενώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν πιο πολυσχηδή εργασία και αυτό αποτελεί μεγάλη ε, πρόκληση και η οικονομική συγκυρία σημαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που ελοχεύουν. Αυτό το είπε και ο Επίτροπος, ο κύριος Μπόρς, γιατί πολλές φορές και οι βιομηχανίες της ε, τροφικής αλυσίδας πρέπει να εξοικονομήσουν, να κάνουν οικονομίες ως προς τους ποιοτικούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας της τροφικής αλυσίδας. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε προβλήματα παρόμοιας φύσης και είναι ενδεικτικό ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο στους ελέγχους ένας από τους δείκτες αφορά την, την οικονομική κατάσταση σε σχέση με τις επιθεωρήσεις. Το μήνυμα είναι σαφές. Εάν η επιχειρήση αντιμετωπίζει οι οικονομικές δυσχέρειες, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν περικοπές στον τομέα της ασφάλειας στην τροφική αλυσίδα. Επίσης, ως προς την πιστοποίηση εξαγωγών. Οι αρχές επιθεώρησης των κρατών μελών θα πρέπει να εξαγάγουν μεγάλες ποσότητες στις τρίτες χώρες και οι έλεγχοι αυτοί θα έπρεπε να διενεργηθούν παντού. Η Λιθουανία μας έδωσε ε, ένα απτό παράδειγμα. Οι Λιθουανικές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν παράλογε απαιτήσει από τις ρωσικέ αρχές, τις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Γι' αυτό θα πρέπει να εξευρεθούν μηχανισμοί έτσι ώστε να προβάλλουμε τα ε, συμφέροντα εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κύριος Πυρίλο μίλησε για την αριστεία όλων αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ένα άλλο θέμα το οποίο ε, μας αφορά άμεσα είναι η ελλείψη στους ελέγχους. Τα κράτη-μέλη κάνουν ε, μεγάλες επενδύσεις, γίνονται πολλές ε, επιθεωρήσεις, έλεγχοι, έχουμε δείγματα από τα εργαστήρια στα εργαστήρια τα οποία και αναλύουμε. Συχνά όμως μέσα στα πλαίσια αυτών των ελέγχων βλέπουμε ότι οι έλεγχοι δεν είναι και οι σωστοί. Πολλές φορές ε, προσδίδονται πολύ για την διενέργεια λανθασμένων ελέγχων. Δεν είναι η πραγματική έλεγχη εκείνη που χρειάζονται. Γι' αυτό θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να έχουν μια καλύτερη πλαισίωση έτσι ώστε να μπορέσουν να στοχοθετήσουν καλύτερα τους πόρους, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για τους σωστούς ελέγχους. Ως προς τις κυρώσεις ο συνάδελφος αναφέρθηκε σε αυτό, δεν θα μπω σε λεπτομερίες, με μία εξαίρεση. Πολύ συχνά ακούμε και προβάλλονται αιτήματα για πιο αυστηρές κυρώσεις. Και αυτό ιδιαίτερα στο σκάνδαλο του αλογίσου κρέατος, όπου ε, αναλύθηκαν πολλοί κίνδυνοι, γνωρίζοντας ότι βεβαίως εάν πιάσουμε τους παραβάτες θα είχαν να υποστούν σοβαρές ε, κυρώσεις. Θα πρέπει όμως να υπάρξει μία σωστή ε, ισορροπία. Θα πρέπει να είναι αναλογικές οι κυρώσεις, γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη πολλές φορές οι κυρώσεις είναι δυσανάλογες και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο για τις αρχές επιθεώρησης να παραπέμψουν μία υπόθεση ε, στο δικαστήριο και πολλές φορές αν είναι δυσανάλογες οι κυρώσεις, οι δικαστικές αρχές ακολουθούν μια αυστηρή γραμμή και αποκλείουν την υπόθεση και αυτό δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε και με ένα θέμα δεοντολογίας όσον αφορά τους ελέγχους αυτούς. Ε, θέματα οργάνωσης καθαρά δυνάμει της πρότασης της Επιτροπής καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε μια σωστή χρηματοδότηση ε, των κρατών μελών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο έργο τους. Αλλά εάν δεν υπάρχει ένας αποδοτικός έλεγχος, τότε όποιες, όποιοι και να είναι οι πόροι και οι προσπάθειες και οι κοινέ προσπάθειες δεν θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, μια σωστή διάρθρωση, διότι στις επιθεωρήσεις βλέπουμε ότι υπάρχει κάκιστη οργάνωση. Δεν υπάρχουν σωστά επίπεδα επικοινωνίας μεταξύ ομοσπονδιακών ε, και περιφερειακών αρχών ή περιφερειακών και τοπικών αρχών. Μπορούμε να μεταβούμε σε ένα κράτος μέλος και να βλέπουμε ε, έναν έλεγχο ex post όπου ε, είχαμε διενέργεια πολλαπλών ελέγχων. Όμως σε ένα άλλο σημείο βλέπουμε ότι υπάρχουν λίγοι έλεγχοι. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται νέα ή ε, νέα κατανομή καλύτερα των πόρων, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σωστά οι πόροι εκεί όπου χρειάζονται. Μία άλλη πρόκληση, η οποία σχετίζεται με το σκάνδαλο στο αλογίσιο κρέας, αφορά τις απάτες και θέματα ποιοτικών ελέγχων. Οι αρχές επιθεώρησης εστιάζουν την προσοχή τους σε θέματα ασφάλειας. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος για την χρήση των ε, πόρων και υπάρχει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το τομέα. Όταν έχουμε όμως να κάνουμε με γεωγραφικούς δείκτες, με ποιότητα ή οργανικά ζητήματα, δυστυχώς αυτά τα θέματα που δεν άπτονται της ασφαλείας άμεσα δεν έχουν προτεραιότητα. Και αυτό βεβαίως είναι και κατανοητό, διότι η ασφάλεια είναι το υπαριθμόν ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε άλλους παράγοντες, γι' αυτό και ο νέος κανονισμός θα πρέπει να εξεύρει τα μέσα μέσα στα πλαίσια των πολιετών προγραμμάτων των κρατών μελών για να γίνεται η σωστή Τώρα, ως προς ε, ειδικού ε, τομείς, ε, όπως ξέρετε στον οριζόντιο τομέα, πολλές φορές δεν υπάρχει ζωστή ανιχνευσιμότητα. Όμως βλέπουμε ότι με το πέρασμα του χρόνου πρέπει να δούμε ορισμένα θέματα που άπτονται των κρατών μελών. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε μεγάλα προβλήματα στα κράτη-μέλη που, όπου ε, υπάρχει θέμα υγειονομικό στο τομέα του κρέατος ως προς τη ε, σήμανση και τα παρασκευάσματα αυτά ε, κρέατος. Επίσης, ως προς τα μαλακόστραγα, ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ως προς τα δίθυρα μαλάκια βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ως προς την ταξινόμηση των περιοχών παραγωγής και ιδιαίτερα ως προς τις τοξίνες, την παρουσία τοξινών. Και γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανταποκριθούν. Ως προς την πρωτογενή παραγωγή, ο Έρικ ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και πρόσφατα βλέπουμε ότι ε, οι διατροφικές κρίσεις, οι κρίσεις ε, τροφίμων δεν έχουν σχέση με ζωικά αλλά με μη ζωικά προϊόντα και ιδιαίτερα στην πρωτογενή παραγωγή. Γι' αυτό οι αρχές επιθεωρήσεων θα πρέπει να προσδώσουν περισσότερο, περισσότερους σπόρους. Και εδώ μιλώ για τρόφιμα και για τα οποροκυπευτικά ιδιαίτερα και τα λαχανικά. Όταν μιλάμε για εισαγωγές, Παραδοσιακά έχουμε ένα πολύ αυστηρό σύστημα ελέγχου ως προς τα ζωικά προϊόντα. Ως προς τα μη ζωικά όμως υπάρχει ένα πιο αδύναμο πλαίσιο, γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν έλεγχο ο οποίος να καλύπτει όλο το φάσμα των προϊόντων. Ως προς την ανιχνευσιμότητα πάντα αποτελεί μείζον πρόβλημα και πρόκληση. Και όπως είπα και ε, νωρίτερα έχουμε περίπου 200 ελέγχους ετησίως τα κράτη-μέλη τα καταφέρνουν πολύ καλά ως προς την εφαρμογή των ελέγχων. Έχει επιτελεστεί μεγάλη ε, ε, πρόοδος τα τελευταία χρόνια και είδαμε ότι ως προς τη σαλμονέλα ε, και μεγάλες ασθένειες στο, στα ζώα έχουν εξαλειφθεί ή έχουν ανοιχνευθεί πρωτίστως. Γι' αυτό προσπαθούμε να ε, βελτιστοποιήσουμε και το πλαίσιο της ανιχνευσιμότητας στο μέτρο του δυνατού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκανέλη, ήταν εκτενέστατη και πολύ εμπεριστατωμένη η αναφορά σας και βάση για την εργασία μας, ότι εκεί ακριβώς θα πρέπει να επέμβουμε όπου υπάρχουν αδιανομίες και ελλείψεις. Χαίρομαι που τηρείτε πάνω κάτω όλοι το χρόνο σας και ελπίζω και οι υπόλοιποι. Και τώρα πάμε στις ανεπάρκειες στη σημερινή νομοθεσία και ανάγκη για έμπρακτε βελτιώσει. Ο Δόκτωρ Μάρτιν Χάρτμαν, αξιότιμε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να σας παρουσιάσω την εθνική ε, οπτική των ε, αρμοδίων επιτόπου στην κάθε χώρα μέλος. Επιτρέψτε μου σύντομα να σας παρουσιάσω τον Γερμανικό Σύλλογο Επισήμων ε, Κτηνιάτρων. Είναι μια δευτεροβάθμια οργάνωση από τα 16 κράτη, τα κρατήδια και εκπροσωπεί πάνω από 5.500 ε, κτηνιάτρους που εργάζονται στο δημόσιο ε, γυναίκες και άνδρες. Και συμμετέχει και στην ΙΑΣΦΟ ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Οργάνωση ε, και στην Ομοσπονδία των Κτηνιάτρων Πανευρωπαϊκά. Με τι ασχολούμαστε. Κυρίως με τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την προστασία των ζώων. One Health. Μία ενιαία είναι η υγεία ανθρώπων και ζώων. Αυτή είναι η σύγχρονη έννοια. Και η ασφάλεια έχει να κάνει από το χωράφι στο ράφι ή από το στάβλο στο τραπέζι μας. Και βασικά έχω να σας πω το εξή για την σημερινή ασφάλεια τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι σαφέστατο η ασφάλεια τροφίμων και η ποιότητα των τροφίμων στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, φτάσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Παρόλα αυτά, δεν ε, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε αποτελμάτωση ή να ευσυχαστούμε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση βάσει νέων καταστάσεων και βάσει νέων εξελίξεων. Θα πρέπει να αντιδρούμε. Και γι' αυτό χαιρετίζω και καλωσορίζω τη μεταξέλιξη του κοινοτικού ε, δικαίου για την αντικατάσταση του κανονισμού του 882 του 2004. Δεν θα αναφερθώ στα θετικά, θα περιοριστώ μόνο σε ορισμένες ανεπάρκειες ε, και ερωτήσεις, υποδείξεις, ε, προτάσεις για τη βελτίωση του ε, σχεδίου. Στο άρθρο 7 αναφέρεται και ο επίσημος έλεγχος και η διαφάνειά του και στόχος είναι η ενιαία υποχρέωση για ενημέρωση ε, των επισήμων ελέγχων. Θα πρέπει πάντα εκεί να γίνεται ε, μια στάθμιση ε, μεταξύ του συμφέροντος των καταναλωτών που πρέπει να προστατεύεται και των εταιριών η Γερμανία έχει αυτό το εργαλείο με την ενημέρωση της κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια ε, και πρέπει να είναι πάρα πολύ γερή η νομική βάση για να αποφύγουμε προβλήματα στην εφαρμογή. Στο άρθρο 7, ε, παράγραφος 3, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αντιτίθεται με το απόρριτο και την προστασία των ε, εμπορικών ε, πληροφοριών αν ενημερώνεται το κοινό για τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνονται οι έλεγχοι. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι αυτό που ανησυχεί τους καταναλωτές και τους αναστατώνει δεν είναι μόνο ε, πληροφορίες ε, για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά ανησυχούν γενικότερα για τις μεθόδους παραγωγής. Ανησύχησαν για το ε, αλογίσιο κρέας πρόσφατα ή για διάφορα σάπια κρέατα που εμφανίστηκαν σκάνδαλα στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε παραπλανητική πληροφόρηση, εξαπάτηση και κανονική απάτη. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 15 για τους επίσημους ελέγχους στην παραγωγή ε, προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Από την άποψή μας ε, παραμένουν κάποια εκκρεμή ζητήματα. Παράγραφος 1 στο άρθρο 15 γενικά αναφέρει τις επίσημους ελέγχους. Ε, θα πρέπει αυτό να συγκεκριμενοποιηθεί ε, στον επόμενο κανονισμό και με βάση τον 853 του 2004 γιατί ακόμα αυτό εκρεμεί και δεν είναι σαφές. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση επισήμων ελέγχων. Η κρεοσκόπηση είναι στοιχείο αυτών των επισήμων ελέγχων και παραμένει επιπλέον. Ο έλεγχος θα γίνεται από επίσημο δημόσιο κτηνίατρο κρεοσκόπο. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ερμηνείας εκεί που μπορεί ε, να οδηγήσει σε παρερμηνείες και να ξεχυλώσει ας πούμε ο ορισμός και η ερμηνεία και χρειάζεται διευκρίνηση. Στη συνέχεια, ε, τι γίνεται με τους ελέγχους, τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Πάντα αναφέρομαι σε ζωικά προϊόντα και ζώα. Ε, αυτά είναι στα άρθρα 53 ε, και 47. Κατά την άποψή μας δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά αυτά. Γίνεται λόγος για φυσικούς ελέγχους των ζώων που θα πρέπει να γίνονται αυτά από δημοσίους κτηνιάτρους. Σωστό είναι αυτό και καλό. Αλλά τι θα πει φυσικός έλεγχος για τα ζώα, ναι, αλλά για τα ε, ζωικά προϊόντα λέει γίνεται από προσωπικό που έχει αντίστοιχη κατάρτιση. Δηλαδή, δεν θα είναι κτηνίατροι αυτοί. Τι ορισμός είναι αυτός. Αυτό το προσωπικό μπορεί να είναι ευρύτερο. Ε, μα όταν πρόκειται για τα ζώα, ε, είναι οι ελεκτές κτηνίατροι, αλλά και τα ζωικά προϊόντα θα πρέπει να ελέγχονται ως προς τις ε, επιζωτίες και την προστασία των ζώων. Και γι' αυτό σαφέστατα θα πρέπει κάποιος να είναι κτηνίατρος για να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Επίσης θα ήθελα να πω ε, όταν δίνονται πιστοποιητικά υγείας για τα ζώα ή και πιστοποιητικά ασφάλειας και υγιεινής, ε, ε, τα ζωικά προϊόντα θα πρέπει να υπογράφονται από κτηνίατρο και στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν πάντα και στα δύο, και στα ζώα αλλά και στα ζωικά προϊόντα να επιφορτίζεται κτηνίατρος πάντοτε με τον έλεγχο αυτό. Χρηματοδότηση των ελέγχων από ε, υποχρεωτικά τέλη. Το ακούσαμε προηγουμένως. Είναι ένα θέμα καθόδες αυτό. Ο στόχος ποιος είναι. να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και να είναι ενιαία και συγκρίσιμη μέθοδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κατά τη δική μας ε, γνώμη, το σύστημα που ισχύει μέχρι τώρα, η δυνατότητα επιβολής τελών δεν είναι κακό. Ε, το έχουμε αυτό στο κρέα, στο γάλα και σε άλλα ζωικά προϊόντα, είναι υποχρεωτικά τα τέλη, αλλά ε, κάποιοι κανόνες για προαιρετικούς ελέγχους θα μπορούσε ε, να γίνει προαιρετική επιβολή τελών, δηλαδή θα μπορούσε ε, να γίνει χωρίς να επιβληθεί αυτό παντού στα κράτη-μέλη. Η καταποκοπή επιβολή τελών νομίζω είναι προβληματική ή δύσκολη για λόγους νομικούς να εφαρμοστεί ενιαία τέλη παντού. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι προδιαγραφές να είναι σαφείς και τα προοπιτούμενα για τον, την επιβολή αυτών των τελών. Με χαμηλό όσο γίνεται διοικητικό κόστος. Θυμίζω τα τέλη που είχαν επιβληθεί για την υγιεινή του κρέατος. Να μην καταλήξουμε τώρα στα δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. εξαίρεση τώρα και απαλλαγή από τα τέλη, το άρθρο 82 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό έχει να κάνει με το διοικητικό φόρτο που δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τις μικροεπιχειρήσεις, πολύ μικρές εταιρείες. Πώς ορίζονται αυτές, κάτω από 10 εργαζόμενοι και κάτω από ετήσιο κύκλο εργασιών 2 ε, ε, εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία αυτό θα αφορούσε 80 με 90% των επιχειρήσεων. Οπότε είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για το πώς θα χρηματοδοτείται ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται. Ιδιαίτερα θα έχουμε μεγάλα προβλήματα και απώλεια εσόδων ε, στους ελέγχους που γίνονται στα σφαγεία που μέχρι τώρα ε, χρηματοδοτούνται από τέλη που πληρώνουν οι ίδιες εταιρείες. Άρα θα μειωθούν τα έσοδά μας και παρόλα αυτά θα πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των ελέγχων που χρηματοδοτούνται από αυτά τα λιγότερα έξοδα. Επίσης, είναι δύσκολο να δούμε, να ελέγχουμε αυτά τα κριτήρια. Θα ζητάμε τη φορολογική δήλωση, δηλαδή από κάθε εταιρεία, αν βγάζει λιγότερα από 2 εκατομμύρια το χρόνο. Και ε, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, που ε, σπάνε σε θηγατρικές ή που ε, αποσπούν προσωπικό και το απασχολούν κάπου αλλού. Έχει παραθυράκια εδώ αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα αν εξαιρούνται οι πολύ μικρέ επιχειρήσει. Αυξάνεται η χρηματοδότηση από το δημόσιο κορβανά αντί να μειώνεται. Και τώρα που είναι τα ταμεία άδεια, όπως έχουμε ακούσει, τα κρατικά, είναι δύσκολο η επίσημη έλεγχη να χρηματοδοτούνται επαρκώς από το κράτος. Οπότε υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε αηφόρους ελέγχους και να μην είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια της ε, τροφικής αλυσίδας. Είναι διακυβευτή. Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαριστεί στο άρθρο 84 είναι ότι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτουν το επιπλέον κόστος και να είναι αυτό υποχρεωτικό. Μπορούμε να βάλουμε όρια, αν θέλετε, κάτω από τα ε, από ένα ποσό ότι θα ήταν πολύ υπερβολικό το κόστος επιβολής του τέλους ε, και το γραφειοκρατικό από το ίδιο το τέλος. Οπότε θα πρέπει να εξαιρούνται. Βέβαια υπάρχουν και μεγάλες επιφυράξεις ε, για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις που θα έχουν σημαντικές λεπτομέρειες για τεχνικά ζητήματα. Και δεν μπορεί τίποτα οριστικό από τώρα να υποθεί. Θέλω να σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, δόκτωρα Χάρτμαν. Σαφέστατες οι απόψεις σας και οι προτάσεις σας. Έχουν ε, υποθεί πολλά. Άλλοι μιλήσατε για τα οικονομικά. Κύριε Μπορέλο, τώρα θα μας μιλήσετε εσείς για τη χρηματοδότηση των επισήμων ελέγχων, για την οργάνωση του συστήματος τελών. Να κάνετε τις δικές σας προτάσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για να σας δώσουμε τη θέση των αρμοδίων αρχών σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι εθνικοί έλεγχοι. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι εκτιμούμε την προσπάθεια της Κομισιόν για την προσπάθεια που κάνει με αυτή την πρόταση κανονισμού. Θέλει να δημιουργήσει μια, ένα πλουστευμένο πλαίσιο επίσημων ελέγχων. Θεωρώ ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα χρηματοδότησης είναι η εκ κάνευ προϋπόθεση για να φτάσουμε σε αποτελεσματικούς ελέγχους που θα εξασφαλίσουν ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, αλλά και των φυτών. Αλλά και θα είναι και προς όφελος των επιχειρηματιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη για το, τα τέλη που εισπράττουν τα κράτη-μέλη για να καλύψουν το γενικό κόστος των γενικών ελέγχων που όπως θυμάστε ε, προτάθηκε από την Κομισιόν, ε, έγινε μάλλον από την Κομισιόν 2009, ε, έγινε ούτως ώστε να βρούμε τους απαραίτητους πόρους μέσα στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Και όμως ο στόχος ο οποίος είχε καθοριστεί για όλα τα κράτη-μέλη δεν έχει υλοποιηθεί και αυτό το υπενθύμησε πριν από λίγο ο συνάδελφος. Οι νέε διατάξεις όμως, κατά την άποψή μου, δεν είναι αποτελεσματικές για να λύσουν τα προβλήματα του συστήματος όπως είχαν εντοπιστεί. Και μάλιστα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη βιωσιμότητα ολόκληρου του συστήματος και να αυξήσουν βεβαίως την δυσαρμονή, μια, αρμονική εφαρμογή των επίσημων ελέγχων. Θα αυξήσουν δηλαδή τη δυσαρμονία αυτή που υπάρχει. Θα ήθελα να κάνω μια γενική σκέψη, ένα γενικό προβληματισμό. Η βασική σκέψη είναι ότι το κόστος της δραστηριότητα του ελέγχου θα πρέπει να βαραίνει τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες με βάση τον, τον παράγοντα του κινδύνου και κατά την άποψή μου ότι αυτή η ιδέα δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι μιλάμε ε, για υγειονομικούς ελέγχους καταρχάς. Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται και για την προσόφελος του, των επιχειρηματιών του κλάδου, που χάρη στη δραστηριότητα του ελέγχου και στη δραστηριότητα της ε, δημόσιας πιστοποίησης μπορούν να βάζουν στην αγορά τα προϊόντα τους όμως αυτές οι ελεγκτικές δραστηριότητες γίνονται και προς όφελος του κοινού καλού ε, για να προβλέψουμε, να προλάβουμε ασθένειες και να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, να την προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Επομένως το κόστος του ελέγχου θα πρέπει να κατανεμηθεί με κάποιον τρόπο και θα δούμε πώς στην συνεχεία μεταξύ των επιχειρηματιών αυτών αλλά και του δημοσίου τομέα δυνάμει των διαφόρων στόχων που προωθούνται. Για την κάλυψη ε, του κόστους των ελέγχων και την προστασία της δημόσιας υγείας, τα κράτη-μέλη θα έπρεπε επίσης να συνεισφέρουν τουλάχιστον μέσω ενός ποσοστού, ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, διάφορες μορφές και να αφήσουμε να πληρώνουν εξ ολοκλήρου τους ελέγχους που γίνονται προς όφελος των ιδιωτών, προς όφελος των επιχειρηματιών. Αυτό είναι το ένα σημείο που ήθελα να πω. Και κάτι άλλο που θα ήθελα επίσης να θίξω, γιατί αναφέρθηκε από προηγούμενους ομιλητές, είναι ότι συχνά ε, τα τέλη που καταβάλουν επιχειρηματίες δεν ε, χρησιμοποιούνται σωστά από τις ε, δημόσιες αρχές. Δεν γίνεται σωστή κατανομή ούτως ώστε θα πρέπει, θα πρέπει να κάνουμε μία αναπροσαρμογή του κειμένου, τόσο ώστε όλα τα ποσά που εισπράττονται να χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους. Κατά την άποψή μου, για να ξεπεράσουμε τα όρια και τους περιορισμούς του σημερινού συστήματος α, χρηματοδότησης, θα πρέπει καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εντοπίσουμε κάποια ενιαία στάνταρ, κάποια ενιαία πρότυπα ε, επίσημων ελέγχων και να καθορίσουμε μία ελάχιστη συχνότητα για όλες τις δραστηριότητες που υποβάλλονται σε έλεγχο με βάση μια, με βάση μια εναρμονισμένη ταξινόμηση του κινδύνου. Η πρόταση κανονισμού προβλέπει ότι η Κομισιόν με μετέπειτα κατεξουδότηση πράξης θα καθορίσει αυτή την ελάχιστη συχνότητα των ελέγχων. Αλλά αυτό είναι μία πρόβλεψη και αφορά μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Σήμερα ξέρουμε και το υπενθύμισε ο προηγούμενος ομιλητής ότι και τα φυτά επηρεάζουν αρνητικά μερικές φορές την υγεία. Παραδείγματος χάρη το, η περίπτωση του κολοβακτηριδίου υπενθυμήθηκε. Ε, επίσης περιπτώσεις υπατήτηδας α που α, είχαμε κρούσματα υπατήτηδας α γιατί κάποια άτομα κατανάλωσαν φρούτα του δάσους τα οποία είχαν μικρόβιο. Όλα αυτοί, όλοι αυτοί οι κινδύνοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν κατά τους κινδύνους. Επομένως θα πρέπει να τυποποιηθούν η έλεγχοι, να υπάρχει μια ελάχιστη συχνότητα και αυτό θα είναι ε, κάτι που θα πρέπει να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο με μια απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου χωρίς αυτό να το αφήσουμε δηλαδή στις κατεξιοδότηση πράξεις της Κομισιόν σε μεταγενέστερες δευτερογενείς πράξεις μέσα σε ένα όριστο χρονικό πλαίσιο. Όχι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να επανέλθω λοιπόν στα υποχρεωτικά τέλη που θα πληρώνουν οι επιχειρηματίε για να καλύπτεται το κόστο του ελέγχου. Η πρόταση κανονισμού δεν προβλέπει τον ορισμό ελάχιστων ενιαίων ποσών. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα βήμα προς τα πίσω σε σχέση με τη σημερινή νομοθεσία. Έχουμε, λέμε δηλαδή ότι τα υποχρεωτικά τέλη αυτή θα καθορίζονται κατά αποκοπή με βάση το κόστος ε, του ελέγχου, ε, όπως το καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο, εξάρτητα ε, αφήνουμε δηλαδή ε, στα κράτη-μέλη τη συχνότητα των ελέγχων, αφήνουμε το, πώς, το ποιος θα ελέγχεται κτλ. Έτσι όμως ε, υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Μπορεί τα κράτη-μέλη να μην έχουν σίγουρους πόρους και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις ε, στην, ε, στην προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του ελέγχου και στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργούν οι αρχές. Γι' αυτό το σημείο προτείνουμε να επανεισάγουμε εναρμονισμένα ελάχιστα ποσά ε, που θα προέρχονται από υποχρεωτικά τέλη, ενδεχομένως ρυθμιζόμενα στα διάφορα κρατημέλη, ανάλογα με παραμέτρους οικονομικοκοινωνικές ε, που θα, θα κρίνουμε απαραίτητε, ούτω ώστε να υλοποιήσουμε το στόχο της ίσης μεταχείρισης των επιχειρηματιών. Ε, θα ήθελα τώρα να σταθώ στο θέμα των μικροεπιχειρήσεων, ευαίσθητο θέμα, λεπτό, το ξέρω πολύ καλά και ξέρω ότι μπορεί να δημιουργήσω και μερικές έκφρασεις θεωρώ ότι αυτή η πρόβλεψη μπορεί να είναι προβληματική για μια χώρα όπως η Ιταλία, όπου το 93% των επιχειρήσεων στο γεωργοδιατροφικό τομέα ε, ταξινομούνται ως μικροεπιχειρήσεις. Από πού θα βρούμε τα λεφτά? Μπορούν τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσουν αυτούς τους ελέγχους που παλιά γίνονταν όταν αυξάνονται κατά 93% ο βαθμός των ε, ελέγχων, ο αριθμός των ελέγχων. Αυτό είναι ερωτηματικό που θέτω. Εμείς θα θέλαμε μέτρα τα οποία ε, βεβαίως να είναι προς όφελος των μικρών παραγωγικών μονάδων, αλλά θεωρούμε πιο δίκαιο και πιο σωστό να προβλέψουμε μια κλιμάκωση του ποσού ε, συνεισφοράς με βάση την πραγματική παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης. Αυτό εμείς το κάναμε στο σημερινό κανονισμό 882. Όλα τα επιχειρήματα που ακούσαμε μέχρι στιγμής ισχύουν ακόμα περισσότερο για τη χρηματοδότηση ε, ελεγκτικών δραστηριοτήτων κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Σε ένα σύστημα όπου ένα εμπόρευμα το οποίο εισάγεται μπορεί να ελεγχθεί σε οποιοδήποτε από τα φυλάκια συνοριακών ελέγχων των 28 κρατών μελών και η συνεχεία μπορεί να απελευθερωθεί στην ενία αγορά, είναι απαραίτητο σαν τέτοιο σύστημα να εναρμονίσουμε ε, του, τα ελάχιστα τέλη που καθορίζουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο ποσοστό, ε, τα τέλη να είναι κάποιο ποσοστό των ε, δασ, δασμών που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το χάρη. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η εναρμόνιση, θα έχει ε, επίπτωση στις εμπορικές ροές. Μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην κοινή στρατηγική βιοασφάλεια στα σύνορα που θέλουμε να εξασφαλίσουμε με το, πρώτο, σχέδιο του προγράμματος παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο το 2007. Συμπερασματικά, θέλω να ξανασκεφτούμε κάποια σημεία του συστήματος χρηματοδότησης των επίσημων ελέγχων όπως προτείνεται από τον κανονισμό, για να εξασφαλίσουμε τους στόχους μας και να περάσουμε σε, εναρμονισμένους, σε εναρμονισμένα επίπεδα τελών, ούτω ώστε να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ και ήταν πραγματική τιμή που μου δώσατε το λόγο για να παρουσιάσω τη θέση μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε και θα μας απασχολήσουν ε, πολύ καιρό ακόμα οι προτάσεις σας. Έχουν πολύ ουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επισκόπηση νέων δράσεων έμπρακτης εφαρμογής και μέτρων κατά της απάτης και παρακαλώ τον κύριο Τζον Μπάρνς να λάβει το λόγο. Thank you very much, Chair, and thank you for inviting me. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω σήμερα ενώπιον σας. Θα ήθελα να σας δώσω μια συνολική εικόνα για τη νέα πρόταση ε, εφαρμογή του πλαισίου για τον τρόπο ε, θέσεως εφαρμογή του πλαισίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πάνω από 400 αρχές εφαρμογή αυτού του πλαισίου που εφαρμόζουν τον κανονισμό 882. Καλύπτουν 600.000 επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών και ε, πρόκειται για περίπου 400-500.000 φορείς στα είδη εστίασης. Έχουμε 100.000 ελέγχους ετησίως που καλύπτονται από τον 882 και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πλαίσιο λειτουργίας. Δίνουμε προτεραιότητα το, στην ασφάλεια τροφίμων. 400.000 έλεγχοι σχετίζονται με αυτό το ζήτημα και αφορούν τη σύνθεση, τη σύσταση και την σήμανση. Ο μόνος λόγος ε, που αναφέρω αυτά τα στοιχεία είναι διότι αποτελούν ένα πολύ καλό τεστ αντοχής στον κανονισμό και πιστεύουμε ότι 882 που αφορά τους ελέγχους τροφίμων και ζωοτροφών μας δίνει ένα συνεπές πλαίσιο το οποίο μας βοηθά για την πραγματική θέση σε εφαρμογή και κατανόηση του πλαισίου. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ευρεία κατανόηση από τους εθνικούς ρυθμιστές, από τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς ρυθμιστές και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Θέλουμε να προωθήσουμε τον παρόντα κανονισμό διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής σε όλη την ε, διατροφική αλυσίδα και αυτό το υποστηρίζουμε καθώς και τα νέα μέτρα που ενυπάρχουν έτσι ώστε να βλέπουμε τι γίνεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, δηλαδή απάτης στα κράτη-μέλη και όπως ξέρετε η βιομηχανία τροφίμων ε, είναι ένας βασικός τομέας και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή είναι ύψης της ε, σημασίας έτσι ώστε να έχουμε μια, έναν καλύτερο κανονισμό, καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού. Η πείρα μας, δυνάμει του 882, σχετίζεται με τις ε, βασικότερες πτυχές του συστήματος. Δεν θα καλύψω το χρηματοοικονομικό, αλλά τη δυνατότητα να στοχοθετήσουμε την πηγή κινδύνων. Είναι μια πολύ βασική συνιστόσα και θα θέλαμε να επεκταθεί. Τώρα μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό θέλουν και οι καταναλωτές, αλλά επιτρέπει στις τοπικές αρχές και στους ρυθμιστές να προβούν σε μια επιμέρους στοχοθέτηση και να δώσουν πόρους στις, ε, στοχοδετώντας μεγαλύτερες προτεραιότητες. Θεωρούμε λοιπόν ότι με βάση τις τρέχουσες προτάσεις και με βάση και τις νέες ε, δυνάμει του 882 θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ήδη η έλεγχη από τις επιχειρήσεις είναι ύψης της σημασίας. Θεωρούμε ότι αυτό ενθαρρύνει την συμμόρφωση της βιομηχανίας η οποία αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Επιτρέπει στους ρυθμιστές και στις τοπικές αρχές στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου να προβούν σε μια στοχοθέτηση με βάση των κινδύνων και τη μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και έτσι επεκτείνουμε αυτές τις προτάσεις για να μιλήσουμε για τα λιμάνια και τη, τους ελέγχους στην ενδοχώρα, κάτι το οποίο θα υποστηρίξουμε. Επίσης, με βάση τον κανονισμό 882, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον τρόπο παροχής εγγυήσεων. Αυτό είναι ύψης της σημασίας όταν μιλάμε για νέους αναδιόμενους κινδύνους. Θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές και στους υπευθύνους έτσι ώστε να αντιδράσουμε τάχιστα στην περίπτωση νέων κινδύνων ή στην περίπτωση του αλογίσιου κρέατος. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις που θα συνεχίσουν να διανοίγουν αυτή την οδό έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ελέγχουν τις παραδόσεις και θα υποστηρίξουμε και την εργασία της ΦΑΟ έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστοι δυνατοί Έλεγχη, γιατί εμείς είμαστε ο πλέον αδύναμος ε, κρίκος στην, στον έλεγχο ποιότητας και σε επίπεδο ελέγχου εργαστηρίων θεωρούμε ότι αυτή η πιστοποίηση καταδεικνύει ότι τα επίσημα εργαστήρια θα μας δώσουν αποτελέσματα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη. υποστηρίζουμε τις προθυμένες προτάσεις, τις ενισχυμένες προτάσεις για μεγαλύτερη ε, διαφάνεια. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες και από τα κράτη-μέλη και από τη βιομηχανία. Οι προτάσεις ε, εισαγάγουν μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ αρμοδίων αρχών και οικονομικών φορέων, καθώς και αρμοδίων αρχών και κοινού εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ένα σύστημα βαθμολόγησης το οποίο ε, διατίθεται και online για όλες τις επιχειρήσεις καλύπτοντας 440.000 επιχειρήσεις. Έτσι οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν που θα ε, λάβουν πληροφορίες σε σχέση με τις προδιαγραφές υγείας και υγιεινής. Εάν θέλουμε ε, να δώσουμε περισσότερη και καλύτερη βαθμολόγηση, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για ένα απλό ε, πλαίσιο και άμεσα προσβάσιμο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει συμμόρφωση και από τότε που έχουμε εισαγάγει αυτό το σύστημα βαθμολόγησης βλέπουμε ότι οι καταναλωτές και η βιομηχανία μπορούν να επιλέξουν με απόλυτη εμπιστοσύνη το προϊόν που επιθυμούν. Επίσης θεωρούμε ότι οι εισηγήσεις της επιχειρήσης είναι, άμεση, είναι άμεσου αποτελέσματος και θεωρούμε ότι αυτό βοηθά στην κατανόηση της ε, λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι και κάτι που αποτελεί πρόκληση, γι' αυτό θα πρέπει οι αρμόδιοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν και αυτό είναι μια βασική ε, συνιστός, ένα βασικό στοιχείο που θα πρέπει να προωθήσουμε στις νέες προτάσεις Επίσης, όπως ακούσαμε και προγενέστερα, θα πρέπει να υπάρχει η εναρμόνιση και απλούστευση στην τροφική αλυσίδα. Ε, αυτό βεβαίως συμπεριλαμβάνει και τις περιοχές των συνόρων, έτσι ώστε να μεταφέρουμε τους σπόρους εκεί που χρειάζονται και να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης από τις επιχειρήσεις και τους ρυθμιστές. Υποστηρίζουμε λοιπόν οποιοδήποτε σύστημα το οποίο ε, μειώνει τη γραφειοκρατία και απλουστεύει το πλαίσιο λειτουργίας. Επίσης υποστηρίζουμε τη νέα ευελιξία στα επίσημα εργαστήρια ελέγχου, διότι πολλές φορές είναι δύσκολο για τους ρυθμιστές να βρουν τη σωστή μεθοδολογία για τους νέους αναδυόμενους κινδύνους που ανακύπτουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να ρυθμίσουμε το πλαίσιο λειτουργίας των επισήμων εργαστηρίων και να υπάρχει και μία ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους νέους αναδιόμενους κινδύνους. Επίσης, δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτικού χαρακτήρα οι προτάσεις ή να έχουν χαρακτήρα αποκλεισμού θα πρέπει να μετρηθούν και με τις μελλοντικές εξελίξεις. Θα πρέπει να κλείσουν οι στότοποι εκεί όπου χρειάζεται και να ε, υπάρχει διοικητική αρρωγή και συνεργασία σε τομείς που δεν μπορούμε καν να εικάσουμε πώς θα είναι. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ε, μειώσουμε τη δυνατότητα ανταπόκρισης. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για τις ενισχυμένες διατάξεις σε σχέση με την απάτη. Πρόσφατα όταν είδα ε, την Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και ε, Ζωοτροφών ε, ξέτασαν ε, μία πίτσα η οποία περιλαμβάνει 25 διαφορετικά συστατικά και πέρασε 60 χώρες και 5 υπήρους. Δεν ήξερα ότι έχει τόσα συστατικά, ούτε ότι περνάει τόσες χώρες. Αλλά βλέπουμε ότι έτσι διευρύνεται και το πλαίσιο ανείχνευσης των, ε, της απάτης. Γι' αυτό χρειάζονται σκόπιμη και καλή έλεγχοι. Στην περίπτωση του αλογίσιου κρέατος υπήρχαν έλεγχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε μία βάση δεδομένων, το Intel του το 12 και δεδομένα από 1380 σημεία. Επίσης, μία, μία βάση δεδομένων και ένα ειδικό ταμείο ε, αντιμετώπισης των κινδύνων. Αυτό όμως που δεν είχαμε ήταν την πληροφόρηση, τη σωστή πληροφόρηση και γι' αυτό υποστηρίζουμε οποιαδήποτε νέα πρόταση που θα μας βοηθήσει στην παράδοση και διάδοση πληροφοριών ανά τα κράτη-μέλη και τη συνεργασία μεταξύ τους. Ε, είναι ζωτική σημασίας για όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Οι νέες ε, διατάξεις για τη μη σκόπιμη ε, μη συμμόρφωση θα πρέπει να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να αντιδρούν όταν υπάρχει ακόμα και υποψία μη συμμόρφωσης έτσι ώστε να έχουμε όλα τα, τα στοιχεία ε, όλα τα στοιχεία μέσω ε, πληροφορικής και επικοινωνιών για να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε την απάτη. Εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν, υπάρχει οικονομικό κέρδος ή υπερκέρδος. Αυτό είναι ένας νέος τομέας και γι' αυτό θα πρέπει να αποθαρρυνθεί αυτό το ε, άλογο κέρδος το οποίο προωθείται από δραστηριότητες απάτης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάνς για τα όσα μας είπατε και αυτά πιστεύω θα μας βοηθήσουν πολύ στο νομοθετικό μας έργο και παρακαλώ τώρα τελευταίο τον κύριο Λοή Κεβέν να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για θέματα εισαγωγών ζώων, ζώντων και ζωικών προϊόντων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, είναι μεγάλη η χαρά και η ευτυχία που έχω να σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Ξέρετε ότι η Γαλλία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις εισαγωγές. Από τον Ιούνιο του 2008 έχει καταθέσει μνημόνιο στο Συμβούλιο που καταλήγει σε συμπεράσματα για τους ενισχυμένους ε, ελέγχους. Λίγο πιο αργά και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να μπορείτε να μεταφράζεστε κιόλας φορές. Euh, D'augmenter να μιλάτε λίγο πιο αργά για να προλαβαίνουν οι διερμηνείς, όχι τίποτα άλλο. Έχω δύο, δέκα λεπτά μόνο, εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η πρόταση γράφεται στη συνέχεια του μνημονίου που είχαμε υποβάλει και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2008 και ε, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας παρουσιάσω ποιες είναι οι βασικές καινοτομίες στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ε, θα σας θυμίσω τι ίσχυε πριν το 2009 για τις εισαγωγές. Βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος παγκόσμιος εισαγωγέας ε, γεωργικών ε, προϊόντων και τροφίμων. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι να ελέγχουμε τι εισέρχεται στην Ένωση. Για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι εξίσου ασφαλές με τα όσα εμείς παράγουμε. Για να προστατεύεται η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων, των φυτών αλλά και του περιβάλλοντος. Τι ελέγχουμε τέσσερις μεγάλες ενότητες, ε, τα ζώντα ζώα, ζωικά προϊόντα, φυτικά προϊόντα ε, και φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό και λοιπά φυτά όπως είναι τα φρούτα. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες φάσεις ε, στην ε, ανάντη φάση στη ζωική παραγωγή η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τι ισχύει στη κάθε χώρα ως προσέλεγχο και έχει και ένα κατάλογο τρίτων χωρών ε, και εγκεκριμένων, εξουδοτημένων ή απαγορευμένων επιχειρήσεων για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνοντας στα σύνορα, τα προϊόντα ελέγχονται φυσικά. Πρώτα ελέγχονται τα παραστατικά. Υπάρχει το υγειονομικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι η εξαγόμενη παρτίδα ανταποκρίνεται ε, στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται και τυχαίος έλεγχος και ε, μέσω των διαφόρων ε, τρόπων που έχουμε για να ελέγχουμε τους κινδύνους του, είτε είναι αυτή η βιολογική είτε είναι χημική. Οι άλλοι έλεγχοι που δεν γίνονται στα σύνορα αλλά γίνονται στον προορισμό όταν φτάνουν τα τρόφιμα και είναι αυτό το τμήμα 1 αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα και τα φυτά που δεν υφίστανται τον φυτογειονομικό έλεγχο. Για παράδειγμα, ε, η έρευνα που γίνεται και ο έλεγχος για τα κατάλοιπα. Α, δυσκολεύομαι με το μηχάνημα. Ε, ο έλεγχος των εισαγωγών βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί εμπορικό εμπόδιο. Γι' αυτό Υπάρχει μια διεθνή συμφωνία και στα πλαίσια του ΠΟΕ που τα ρυθμίζει αυτά. Το δόγμα είναι απλό. Οι φραγμοί όταν μπαίνει σε μια χώρα επιτρέπονται και τα εμπόδια όταν δικαιολογούνται και από τι δικαιολογούνται από τους διεθνείς κανόνες. Είναι τρία τα όργανα αυτά, ο Κόντεξ Alimentarius, ε, το Διεθνές Γραφείο Επιζωτιών και ο αντίστοιχο Οργανισμός για τα Φυτά, για τη φυτιο, Υγειονομική Προστασία. Και επίσης υπάρχει και αρχή της ανάλυσης του κινδύνου που επιτρέπει να ε, δικαιολογούνται οι έλεγχοι αυτοί και να επιβάλλονται. Και είναι, φυσικά είναι φραγμός και τροχοπέδι στις εισαγωγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των κρατών μελών της έχει δημιουργήσει ένα ειδικό δίκτυο συνοριακών σταθμών που ειδικεύονται αφενός τους κτηνιατρικούς και φετέρους τους φυτοϊγειονομικούς ελέγχους. Σήμερα είναι διαφορετικές οι απαιτήσει και μία από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υπάρχει ένα ενιαίο σταθμός ε, μεθοριακός για τον έλεγχο που να ανταποκρίνεται σε αντίστοιχες απαιτήσει. Στη Γαλλία εδώ και τρία χρόνια έχουμε ε, και πολλές φορές έχουν συγχωνευτεί οι ε, φυτοϊγειονομικοί με τους κτηνιατρικούς ελέγχους σε μια εθνική υπηρεσία και αυτό έχει πλεονεκτήματα την αμοιβιοποίηση και γίνονται και οικονομίες κλίμακος. Ε, βλέπετε εδώ το χάρτη της Γαλλίας με τους διάφορους μεθοριακούς σταθμούς που είναι ε, λογικά στα αεροδρόμια και στα λιμάνια σύνολων 77 και 87 πλήρους απασχόλησης ε, εργαζομένους και ένα επιτελείο 5 διευθυντών στο Παρίσι. Ε, είναι η έλεγχη βέβαια τελωνιακή και μία από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών αρχών ε, αλλά και των τελωνίων των κρατών μελών. Εναρμόνιση λοιπόν των ελέγχων εισαγωγών στα κτηνιατρικά ε, έχει ε, ένα μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα ενοποιημένο που λέγεται Trust, Trace και επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνονται όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί για μια παρτίδα ελαττωματική η οποία κάπου έχει εντοπιστεί για να μην μπορέσει μέσα από άλλα παραθυράκια να διαφύγει σε άλλο κράτος μέλος. Και υπάρχει και το RAS, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που προειδοποιεί για ε, πιθανώς επικίνδυνα προϊόντα. Έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματικό στην πράξη σε βαθμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στον κανονισμό να διευρυνθεί το ΡΑΣ και να επιβάλλεται σε όλους τους ελέγχους στα σύνορα, όχι μόνο τους κτηνιατρικούς αλλά και τα φυτικά και τις ζωοτροφές. Γίνονται ήδη εμπειρικά τέτοιες δράσει σε κάποιους σταθμού και νομίζουμε ότι αυτό θα αποδώσει και θα αυξηθεί και η αποτελεσματικότητα και η εναρμόνιση. Τώρα, είναι επίσημη αυτή η συνοριακή έλεγχη και είναι αρμοδιότητα του κράτους και πώς χρηματοδοτούνται. Έγινε μεγάλος λόγος προηγουμένως και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί. Ε, χρηματοδοτούνται από τέλη που καταβάλουν οι φορείς ε, του εμπόριου στους αρμοδίους. Προηγουμένως μιλήσαμε για την εξαίρεση από ε, την επιβολή αυτού του τέλους των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αυτό είναι προβληματικό γιατί σήμερα υπάρχουν εταιρείες που καταβάλουν αυτό το τέλος και αύριο θα εξαιρούνται. Άρα μειώνονται τα έσοδα στον προπολογισμό των κρατών μελών και θα πρέπει πολύ προσεκτικά να το μελετήσουμε αυτό. Θα ήθελα να επιμείνω σε ένα σημείο το οποίο προηγουμένως αναφέρθηκε και από τον κύριο Σκάνελ και από τον κύριο Πούλινε σε ό,τι αφορά ε, την εισαγωγή και τις διακρίσεις που γίνονται ανάμεσα στα ζώα και τα φυτά. Υπάρχει ένα σύστημα αδειοδότησης και έγκρισης. Στο ζωικό τομέα τι γίνεται. Είναι κλειστό το σύστημα. Εδώ και πολύ καιρό στην Ευρώπη υπάρχει ένα σύστημα ε, θετικών καταλόγων. Δηλαδή ό,τι δεν αναφέρεται ρητά, ό,τι δεν επιτρέπεται να εισαχθεί, απαγορεύεται. Ε, στο φυτικό κλάδο ισχύουν περίπου τα αντίθετα. Είναι αρνητικό ο κατάλογος, ανοιχτός. Ό,τι δεν απαγορεύεται ρητά, επιτρέπεται να εισάγεται. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι εμπορικοί μα εταίροι και μεγάλες χώρες έχουν κλειστό κατάλογο και για τα φυτά, όχι μόνο για τα ζώα. Άρα εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Δηλαδή, κινδυνεύουμε να προστατευόμαστε λιγότερο καλά ε, από εισαγωγές από κάποιες χώρες οι οποίες μας βάζουν φραγμούς εκείνες για τους ίδιους φυτοϊγειονομικούς λόγους δεν εισάγουν τα δικά μας προϊόντα. Μια στιγμή εδώ υπάρχει κίνδυνος ε, στρέβλωσης και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε. Για να σας εξηγήσω τι εννοώ ως προς την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Βλέπετε στην οθόνη δύο στοιχεία. Στη Γαλλία βλέπουμε ότι έχουμε 3% μη συμμόρφωσης ε, τα τρία τελευταία χρόνια στο φυτικό τομέα, ενώ στο ζωικό ε, είναι κάτω από 1% αυτή η μη συμμόρφωση. Στα φυτά επιπλέον έχουμε μια τεράστια πίεση ε, στον έλεγχο στα σύνορα, γιατί ο έλεγχος αυτός κανονικά θα πρέπει να γίνεται στις χώρες, όχι όταν φτάζει Και το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να ε, είναι στην αρχή και όχι στην, ε, στο τέλος αυτού του δρόμου όταν φτάνουν τα φυτά στην Ένωση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βελτιώνεται η κατάσταση ως προς τις αγωγές τα φυτά μας κινδυνεύουν, τα δάση, ε, οι κήποι, ακόμα και οι λεωφόροι ε, όπου κινδυνεύουν στην Ευρώπη τα δέντρα από ένα παράσιτο, ένα κόκκινο σκαθάρι και θα πρέπει να είναι πραγματικά προληπτική και όχι θεραπευτική η προσέγγιση μας, όπως είναι σήμερα, κυρίως θεραπευτική. Υπάρχει η αντίρρηση ότι το κλειστό σύστημα δεν είναι συμβατό με τον ΠΟΕ. Εγώ ισχυρίζομαι το αντίθετο. Ε, δεν θα πρέπει να γίνει μια διακοπή ξαφνική ε, στους ε, κλάδους που δεν εμφανίζουν κανένα πρόβλημα. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνεται αυτό προοδευτικά και όχι βία και απότομα. Συμπέρασμα. Οι προτάσεις που έγιναν για τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για μας πρόοδος, ε, αλλά στο φυτικό τομέα είναι ανεπαρκής. Τα καταλάβετε άλλωστε από αυτά που σας είπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προστατεύεται από τους εξωτερικούς υγειονομικούς κινδύνους, όπως και οι εμπορικοί της ε, εταίροι το κάνουν και όχι μόνο οι πολύ μεγάλε χώρες, και άλλες χώρες. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει αυτά να τα έχει υπόψη τη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Εβά. Νομίζω ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές τώρα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Κλάς, αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, για να αρχίσει η συζήτηση. Κυρία Λουλάη Άγγι, ευχαριστώ πολύ Χόρσνεχαρτ. και ευχαριστώ και εγώ τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες για τις τοποθετήσεις. Νομίζω ότι πολλά είναι τα σημεία που μπορούμε να συζητήσουμε και ερωτήσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω τη συνάδελφο από τον Καναδά και να της δώσω το λόγο να ανοίξει τη συζήτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μόνο εσωτερική αγορά, είναι και παγκόσμια αγορά στην οποία συμμετέχει και καλό είναι να έχουμε καλή συνεργασία με τις άλλες χώρες, έχει νόημα. Να μας μιλήσετε για τη χώρα σας παρακαλώ, να μας κάνετε την εισαγωγή. Um, Ευχαριστώ που με καλέσατε Διαβάσαμε καταρχάς με μεγάλη προσοχή όλες, όλη την προτινόμενη νομοθεσία σας, όπως υποβλήθηκε μέσω του ΠΟΕ. Και βεβαίως παρακολούθησα και τις παρουσιάσεις σας σήμερα το απόγευμα ε, και πρέπει να σας πω ότι και εμείς είμαστε εν μέσω μεταρρύθμισης της νομοθεσίας μας για τα τρόφιμα και έχουμε μια νέα νομοθεσία, ένα νέο νομοθέτημα στις αρχές του 2013 παρουσιάστηκε, είναι η πράξη ε, ασφαλών τροφίμων για τους Καναδούς. Έχει πολλές ομοιότητες με τη δική σας πρόταση και υπάρχει ευθυγράμμιση σε διάφορα θέματα. Βασιζόμαστε και εμείς στον κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κοινή τάση σε όλες τις προτινόμενες προτάσεις νομοθεσίας και, και η νομοθετική πράξη φύσμα των Αμερικανών, των νότιων γειτόνων μας. Όλη η προσπάθεια εξυγχρονισμού της νομοθεσίας μας, όπως και η δική σας, ε, έχει σαν σκοπό να απλουστεύσει διάφορα νομοθετήματα, να τα εντάξει ένα πλαίσιο, να καταστήσει πιο εύκολο το σύστημα για την ε, βιομηχανία, για τον κλάδο, να αυξήσουμε επίσης ε, τις κυρώσεις για τις απάτες, όπως είπατε και εσείς και προτείνετε και εσείς, να δούμε επίσης και εμείς την ε, χρηματοδότηση του συστήματος. Το σύστημα χρηματοδότησης της ε, ε, υπηρεσίας επιθεώρησης το σύστημα αυτό χρηματοδότηση δεν έχει αλλάξει πότε που δημιουργήθηκε η υπηρεσία το 97 και είναι λίγο απαρχιωμένο. Δεν έχω να σας πω διάφορες λεπτομέρειες για την νομοθεσία, γιατί θα προταθεί την άνοιξη του 2014 και τότε θα σας δώσω λεπτομέρειες. Είμαι ανοιχτή όμως να ακούσω οποιασδήποτε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Υπάρχει μια παρουσίαση από τον Colin Barnes ε, στην ιστοσελίδα μας, την Colin μάλλον. Εκεί μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερες από ό,τι σας είπα εγώ. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πρόκειται για δύο προτάσεις νομοθετικές, η δική μας και η δική σας, που έχουν πολλά κοινά σημεία τελικά. Ε, σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι η γραμματεία έδωσε αυτή την παρουσίαση σε όλους, άρα όλη την εξέταση. Λοιπόν, να σας πω πώς συνηθίζουμε να συζητάμε εδώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους σκιώδης εισηγητές, καταρχάς στο σκιώδης εισηγητή του ΕΛΚ, για να δω αν έχει νέες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε τώρα πολύ γρήγορα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να συγχαρούμε τους υπεύθυνους για την πρόταση. Στην αρχή είχα λίγο τρομοκρατηθεί όταν είδα ότι μας παρουσιάσουν κάτι τόσο περίπλοκο από πλευράς κομισιών, ενώ περιμέναμε μια απλή διόρθωση του πλαισίου. Αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό τελικά να ομαδοποιήσουμε σε ένα κείμενο όλα τα είδη ελέγχων, να ενοποιήσουμε λοιπόν το όλο και να το πλουστεύσουμε. Θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην υπάρχουν πολλοί κανόνες που θα πρέπει να αλλάξουμε συνεχεία. Ελπίζω ότι το κείμενο το οποίο έχουμε τώρα στη διάθεσή μας και το κείμενο το οποίο θα έχουμε για τους κανόνες που θα ακολουθήσουν θα λάβουν υπόψη κάποια πράγματα που υπάρχουν σήμερα. Βεβαίως η κατεξιοδότηση πράξης θα πρέπει να επαληθεύονται, Θα πρέπει να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυ σε ποιο βαθμό αυτές οι κατεξιοδότηση πράξεις επιτρέπουν διευκρινήσεις και σε ποιο βαθμό μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Ένα μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι και η χρηματοδότηση. Έγιναν πάρα πολλές προτάσεις και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εγώ είμαι Γερμανός, τι να κάνουμε και συζητώ ε, με τους αρμοδίους από τη χώρα μου, αρμοδίους για τους ελέγχους και έχω συζητήσει σε διάφορες περιφέρειες και κατατόπους ε, και είναι πολύ μικρέ τελικά οι εταιρείε που θα εξαιρεθούν. Άρα πώ θα χρηματοδοτηθεί αυτή η δράση. Ε, η Γερμανία είναι ένα ομοσπονδιακό κράτο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο αυτό δυστυχώ δεν εφαρμόζεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόβλημα τη χρηματοδότηση. Δεν μπορούν να εξαιρεθούν όλε οι εταιρείε σε κάποιο μέρο. Γιατί είναι η αρμοδιότητα τη τοπική αυτοδιοίκηση και δεν θα έχει καθόλου πόρου. Και στο παρελθόν προσέφηγαν πολύ στο δικαστήριο. Σωστό είναι να λυθεί αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει, αλλά με ποιο τρόπο θα λυθεί. Η σημερινή πρόταση για μένα είναι ανεφάρμοστη. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες ε, <clears throat> προσπάθειες. Το θέμα ε, ε, δεν είναι να ακούτε εμά ως και οδησηγητές, αλλά τι πρέπει να κάνετε εσείς στην πράξη. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ και θέλω να ακούσω εσάς. Ευχαριστώ πολύ Χόρσναχαρτ. Τώρα. Αφήνω τον κύριο Πυρίγιο, τον εισηγητή, να μιλήσει τελευταίος, αν συμφωνεί βέβαια. Ναι, ωραία. Και να δώσω πρώτα το λόγο στον Μπαρτ Στάσκι, ο εισηγητή των Πρασίνων και μετά στην κυρία Γκέρλινγκ και πάει λέγοντας. Λίντα Μακάβαν και λοιπή. Ο Μπαρτ Στάσκι, ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ερωτήσει έχω. Πρώτη, στον εκπρόσωπο του Γραφείου Τροφίμων και το κτηνιατρικό του κυρίου Σκάνα. Ακούσαμε ότι γίνονται πολλές περικοπές στα κράτη-μέλη και αυτό θα επηρεάσει και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η κάθε κρατική αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων. Υποθέτω όμως ότι αυτό επηρεάζει και το δικό σας οργανισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτές οι περικοπές συγκεκριμένα πώς επηρεάζουν τη δική σας λειτουργία στο Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων και στο προσωπικό. Ο κύριος Νέλχαρτ, και έρχομαι στο δεύτερο, μίλησε για τη χρηματοδότηση των ελέγχων και πώς θα γίνει αυτό στο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι κομβικό στοιχείο της συζήτησής μας στην ε, αναδιατύπωση της νομοθεσίας και θέλω να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Πούντελε. Υποθέτω, τουλάχιστον η δική μου θεώρηση είναι ως εξής. σε τελική ανάλυση θα πρέπει να είναι αρμόδιο πάντα το κράτος για τους σωστούς επισήμους ελέγχους. Εντάξει, να είναι ανεξάρτητοι ε, εμπειρογνώμονες που δρούν υπό την προστασία του κράτους, υπό την έγκριση του κράτους, είναι εντεταλμένοι, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του κράτους και να είναι αρκετά αποτελεσματικό. Μπορεί να είναι αυτή η αυτοέλεγχη, οτιδήποτε θέλετε, αλλά τελικά θα πρέπει τη σφραγίδα να τη βάζει το κράτος και να είναι αποτελεσματική έλεγχη και ανεξάρτητη ανεξάρτητη αποκρατική αρχή. Ερώτηση λοιπόν, αν περάσουμε τώρα σε ένα σύστημα που θα καταβάλουν τα τέλη ενδιαφερόμενοι, τα διαβόητα τέλη, για να μην πω τα περίφημα, πώς εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία ε, των ελέγχων. Μπορεί κάποια στιγμή Ακριβώς επειδή οι εταιρείε χρηματοδοτούν ε, τον έλεγχο, μπορεί να επηρεάζουν και το αποτέλεσμά του. Πώς θα βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχει αρνητική επίδραση ε, στον ανεξάρτητο και στον αποτελεσματικό έλεγχο από το κράτος το ίδιο. Μήπως αρχίζουν να παίζουν εκεί οικονομικά κριτήρια ότι α, ας κάνουμε λιγότερους ελέγχους σε κάποιους κλάδους με άλλο τρόπο γιατί δεν έχουμε τα λεφτά εσείς στις προτάσεις σας πώς μπορείτε να εξασφαλίζετε την πλήρη ανεξαρτησία όλων αυτών. Ευχαριστώ Μπαρτσάς και τώρα η Τζο Γκιορλίνγκ αν επιθυμεί πάντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και γι' αυτό θα ήθελα να σταθώ μόνο σε ορισμένα στοιχεία προς τον κύριο Κοντλέ ως προς την ε, βάση, ε, την νομική βάση αυτού του νομοθετήματος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε γιατί είναι αναγκαία η βασική νομοθεσία, τι προσθέτει. Αν τα συμπεριλαμβάνουμε όλα κάτω από ένα τίτλο, δεν ξέρω κατά πόσο ε, υποβοηθούμε κάτι. Αλλά αυτό δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Θα πρέπει να καταδείξουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, θα είναι πιο αποδοτικά. Ποια σκέψη διέπει αυτό το νομοθέτημα. Όταν το δούμε άρθρο προς άρθρο, σε σχέση με τα μετακίνηση των ζώων, ας πούμε για παράδειγμα, εμείς έχουμε δαπανίσει πολύ χρόνο για την ε, μετακίνηση των ζώων. Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες, για όλους μας και σε αυτό το νόμο πλαίσιο ε, αναφέρεται αυτό το θέμα σε πολλά άρθρα. Αλλά στην ουσία ε, περνάμε αυτά τα θέματα χωρίς να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ασχοληθούμε, δηλαδή να αφιερώσουμε τον κατάλληλο ε, χρόνο για να μπορέσουμε να αναφερθούμε σε αυτά τα ζητήματα σε περισσότερη με λεπτομερία. Ε, αν οι μικρές επιχειρήσεις δεν καταβάλουν το αντίτιμο, τότε ποιος θα το καταβάλει. Αυτό αναφέρθηκε, αλλά και το θέμα της επικουρικότητας είναι σημαντικό. Όταν μιλάμε για ένα υποχρεωτικό πλαίσιο δαπανών και καταβολών, ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το γενικεύσουμε. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε το χρόνο για να το δούμε σε αυτό το νομοθετικό έργο. Προς τις κατάλληλες κυρώσεις, και εδώ μπαίνει το θέμα της επικουρικότητας. Αν πρόκειται για ποινικέ διώξεις, πώς μπορούμε να έχουμε ένα νομοθέτημα που να καλύπτει και τα 28 κράτη-μέλη. Νομίζω ότι θα πρέπει βεβαίως να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, πιο κυρωτικό, να γίνονται ποινικέ διώξεις. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν αναλαμβάνεται η κατάλληλη δράση, η επαρκής δράση και αν δεν αναλυφθεί τότε δεν θα καταφέρουμε τίποτα η Λίντα Μακέβαν, και η Σοφιοκονή. Και εγώ άκουσα τους πάντες και είδα τη νομοθεσία στο μεγαλύτερο μέρος της. Ο κύριος Πουτλέ ίσως μπορεί να μας εξηγήσει. Είχαμε δύο μεγάλα σκάνδαλα τροφίμων στη Γερμανία που πέθαναν άνθρωποι τρώγοντας σαλάτα. Δηλαδή αυτά τα Αυτές τις φύτρες ε, λαχανικών. Βεβαίως υπήρξε απάτη στη δεύτερη περίπτωση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η χνηλάτιση των απατών της απάτης για να βγει από το σύστημα. Γιατί αυτό που έχει σημασία άκουσα να γίνεται λόγος για διαφορές μεταξύ των ελέγχων ως προς τα φυτικά προϊόντα σε σχέση με τα ζωικά. Αυτό το ανέφερε και ο Γάλλος συνάδελφος και μίλησα και με την ε, επίσημη αρχή ασφάλειας των τροφίμων στις ΕΠΑ, δηλαδή την ασφάλεια σε όλη την τροφική αλυσίδα, πώς επιλύουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένας θετικός κατάλογος, υπάρχει στην Ευρώπη, γιατί άλλες χώρες δεν τον διαθέτουν. Ως προς τον κύριο Σκάνελ θα ήθελα να μου μιλήσει περισσότερο για ποιοτικά θέματα. Μίλησε για το θέμα της ασφάλειας ε, τροφίμων που είναι τόσο σημαντικό και όχι τόσο η ποιότητα και κάτι άλλο, σε κάτι άλλο αναφέρθηκε. Και Ορισμένοι επιθεωρητές ε, κρεατών είπαν ότι επειδή επήλθαν αλλαγές στο πλαίσιο του 2004 δεν μιλάμε πια τόσο πολύ για ποιότητα. Υπάρχει ένα θέμα ποιότητα στην ε, ε, κατανάλωση κρέατος. Αληθεύει ότι πριν το 2004 η ποιότητα ήταν καλύτερη και τώρα ακολουθεί φθήνουσα απορία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Χάρτμαν μίλησε για τον ε, ρόλο των, ε, της επιθεώρησης από τους ε, κτηνίατρους. Πώς γίνεται ο έλεγχος μεγάλης επιχειρήσης μέσα στα πλαίσια της ρύθμισης. Θεωρείτε ότι η νέα πρόταση εξασφαλίζει τους ανεξάρτητους ελέγχους από κτηνίατρους στον τομέα των, της υγιεινής κρέατος. Μίλησα στον Ηνωμένο Βασίλειο με υπευθύνου ή επιθεωρητές του τομέα του σκανδάλου του αλογίσιου κρέατος, αλλά στο λιανικό εμπόριο εκεί αποστέλλονται άλλοι επιθεωρητές ε, στα, στα μεγάλα ε, εργοστάσια και βλέπουμε δηλαδή ότι γίνεται έλεγχοι αλλά ο λιανικός τομέας δεν μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με το δημόσιο τομέα. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η Επιτροπή. Το είδα ε, και στον τομέα των επιθεωρήσεων. Βλέπουμε δηλαδή τα, τις προδιαγραφές και βλέπουμε ότι οι αγρότες ε, θα ήθελαν να υπάρχει ένα ε, πρότυπο ας πούμε στον, ε, στο τομέα του ελέγχου για τις μπανάνες, να μην υπάρχουν 15 διαφορετικά πρότυπα. Αλλά πολλές φορές γίνονται μεγάλες επιθεωρήσεις, πολλές επιθεωρήσεις στις μεγάλες μονάδες, αλλά όχι στα μικρά σφαγεία. Μου είπαν οι επιθεωρητές ε, κρέατος ότι ένα από τα θέματα ως προς το, στο σκάνδαλο για το αλογίσιο κρέας είναι ότι δεν ε, υπήρχε έλεγχος ε, στα κρέατα, δηλαδή στα σφαγεία. Το θέμα αυτό πώς θα επιληθεί, ιδιαίτερα σε σχέση με τα μικρά σφαγεία, διότι αυτό που έχει σημασία είναι όχι τα μεγάλα σφαγεία, αλλά τα μικρά δηλαδή εκεί που γίνεται η κοπή του κρέατος. Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε στο κοινό. Γιατί χρειάζεται αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση. Ποια είναι τα μικροπαραθυράκια, τι πρέπει να επιλύσουμε και ποια είναι τα χάσματα. Η Σοφία Κονή. Ευχαριστώ πολύ Κρίστα. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω την πρωτοβουλία των συναδέλφων Σνέλχαρτ και Κλάς ε, που διοργανώσατε αυτή την ακρόαση. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά. Σας ευχαριστώ και μπράβο σας γιατί θέτετε τα σωστά ερωτήματα. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στους ελέγχους. Όλοι έχουμε επίγνωση ε, του γεγονότος ότι σήμερα το πρόβλημα είναι ο έλεγχος. Νομοθεσία υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που λείπει είναι ε, το να ελέγχουμε και την προέλευση του κρέατος που μεταποιείται. Αλλά ε, ε, η νομοθεσία είναι καλή και λειτουργική. Το θέμα είναι ο έλεγχος και το πρόβλημα. Εγώ έχω πολλά ερωτήματα. Πρώτον, οι έλεγχοι έχουν τις ίδιες απαιτήσει του ίδιου επίπεδου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέω πλούστατα, διότι κοίταξα κάτι που δεν αφορά τη διατροφή, αλλά ε, τα φυτεύματα μαστού. Στη Γαλλία η εταιρεία που εξαπάτησε εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών με αυτά τα προϊόντα, γιατί το έκανε. Γιατί δεν είναι άδεια να κυκλοφορήσει στη Γαλλία το προϊόν και αυτοί πήγανε ε, σε ένα εξωτερικό εργαστήριο ελεκτικό, δεν θυμάμαι σε κάποια χώρα μέλος, που της έδωσε την έγκριση κυκλοφορία στην αγορά, στη χώρα εκείνη. Ε, στη Γαλλία, στην Ευρώπη λοιπόν, έλεγχοι είναι οι ίδιοι παντού σε όλα τα κρατημέλη. Είναι το ίδιο το επίπεδο των απαιτήσεων. Μήπως θα πρέπει να έχουμε ένα αρμονισμένο έλεγχο παντού σε όλα τα κρατημέλη. Ερώτηση δεύτερη. Για τα αγροδιατροφικά προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το επίπεδο ελέγχου εκεί. Έχω εδώ τον κατάλογο, είναι δεκάδες ε, σελίδων ε, διατροφικών σκανδάλων, ασθενειών και θανάτων ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδέονται με τέτοιου είδους ε, επιδημίες. Και θα αναρωτιέμαι, ο έλεγχος σε κάθε χώρα μέλος είναι ο ίδιος για τις αγωγές μιλώ. Και τρίτον, οι κυρώσεις. Γιατί, εντάξει, καλός ο έλεγχος, αλλά η επιβολή κυρώσεων ποια είναι. Δεν πρόκειται κανείς να εμποδίσει τους απατεώνες να βγάζουν περισσότερα χρήματα εξαπατώντας και με τρόπο ε, παράνομο στα θέματα των τροφίμων. Είδατε τι έγινε με τον κοιμά από κρέας ύπου στο Βόιο. Εκεί τι διαπιστώσαμε. Ο πώς να το πω, ο βιομήχανος αυτός που ε, ήταν στην πηγή του σκανδάλου θα υποστεί μικρότερη τιμωρία από ότι μία νοικοκυρά που έκλεψε δύο-τρεις φορές ένα τρόφιμο για να ταΐσει τα παιδιά της σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Σε αυτήν επιβάλλεται μεγαλύτερη τιμωρία. Λοιπόν, οι ποινές είναι εναρμονισμένες παντού στα κράτη-μέλη και αρκετά μεγάλες για να είναι αποτρεπτικές για τους απαταιώνες για να τερματιστεί αυτή η εγκληματική τους δραστηριότητα. Επόμενη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο με τα φύτρα, τι ήταν αυτό, θυμάστε. Είναι σπόροι που φυτρώνουν. Θυμάστε με την εσερίχια κόλλη, το κολοβακτηρίδιο και είχε και νεκρούς και πολλούς. Μέχρι να μάθουμε την προέλευση, που ήταν γερμανική, από ε, μια γερμανική εκτροφή. Κατηγορήθηκαν οι ε, Ισπανοί ε, παραγωγοί οπωροκυπευτικών, γιατί είχαν πει ότι είναι από αγκούρια που είχαμε εισαγάγει από την Ισπανία και δυσκολεύτηκαν οι άνθρωποι και, και δεν αγόραζαν τα προϊόντα τους γιατί κυκλοφορούσαν διάφορες ανοησίες. Δεν θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφύγουμε αυτή την επικοινωνία που ήταν και λανθασμένη και που προκάλεσε τέτοια προβλήματα και δυσκολίες στα ισπανικά απορροκυπευτικά. Και ένα τελευταίο, αντικειμενικά τώρα. Μια στιγμή πρέπει να τελειώσει, είναι σημαντικό και θέλω απάντηση. Αντικειμενικά, στη Ρουμανία ήξεραν ότι εκατοντάδες ε, είχαν καταλήξει στο σφαγείο ε, γιατί εξελίσσεται η κοινωνία και φύγανε από τα άλογα που τα χρησιμοποιούσαν και τα πήγαν στο σφαγείο και ξέρανε ότι δεν θα φαγωθούν εκεί γιατί δεν αυξήθηκε η κατανάλωση υπείου κρέατος. Και διερωτώ με, στα δικά μας υπουργεία, γεωργίας και τα λοιπά, δεν ξέραμε ότι αυτό το κρέας κάπου θα καταλήξει στην αγορά. Ότι κυκλοφορεί κρέας αλόγου. Μήπως θέλω τη φλήσαμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Και συμφωνώ αυτό για τον έλεγχο. Ρωτάνε και στις δικές μας χώρες οι καταναλωτές. Είναι παντού οι ίδιοι και μήπως να καλέσουμε τους ελεγκτές και τους επιθεωρητές από άλλες χώρες για να κάνουν τους ελέγχους. Εντάξει, πολλές ερωτήσεις. Πολύ σύντομα παρακαλώ, εισηγητής ο κύριος Πυρίλιο, Πυρίλο και μετά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι την ε, Καναδέζα εκπρόσωπο. Στην καναδική νομοθεσία προβλέπετε κάποιες εξαιρέσεις για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Είχατε περιπτώσεις απατών σε τρόφιμα όπως εμείς. Πολύ συγκεκριμένα. Θαυμάσια. Όλοι γνωρίζουν ποιες ερωτήσεις τους έγιναν. Ο κύριος Πούντλε με τη σειρά. Πάρα πολύ γρήγορα να απαντήσετε όλε τι πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει που σας έγιναν. Αδύνατον. Θα πρέπει να απαντήσω ε, πολύ λακωνικά σε κάθε μία από την ερώτηση. Κανονικά έπρεπε να απαντήσω κανένα τέταρτο στην κάθε ερώτηση. Τέλο πάντων, ξεκινάω με σειρά σημασία. Καταρχά με τι κυρώσει. Η Κομισιόν δεν έχει τη δυνατότητα νομικό πώ να εναρμονίσει τι κυρώσει. Δεν μπορεί να πει σε ένα δικαστή 20.000 ας πούμε ε, ευρώ πρόστιμο και 5 μέρες φυλακή στο τάδε άτομο. Όχι, αυτό είναι απόλυτη ευθύνη των κρατών μελών. Αντίθετα σε αυτό το σχέδιο κειμένου έχουμε εκφράσει την επιθυμία μέσω ενός άρθρου οι κυρώσεις, οι χρηματικές κυρώσεις να είναι αναλογικές με το κέρδος του απαταιώνα. Ανάλογα με την απάτη που έκανε. Και θα αποφασίσει βεβαίως τελικά ποιος ο δικαστής υπάρχει μόνο ο προσανατολισμός από πλευράς μας, αλλά και μια μεγάλη ευελιξία συνεχεία που δίδουμε. Για τη χρηματοδότηση τώρα, από τις ε, μικρές ε, επιχειρήσεις ή την εξαίρεση που έχουμε προβλέψει για αυτές. Είναι πολιτικής ε, υφής αυτή η απόφαση. την πήρε για πολιτικούς λόγους, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, για να μην τιμωρήσει τις μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες γενικά παραπονιούνται πολύ για διοικητικά προβλήματα, για διοικητικό άχθος, ε, πολλά έγγραφα που πρέπει να συμπληρώνουν κτλ. και ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορούν να δουλεύουν με λιγότερους ελέγχους από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Προφανώς είναι πολιτικής φύσεως αυτή η απόφαση να τις εξαιρέσουμε και ξέρουμε ότι 80-90% των πελατών των οργανισμών ελέγχου, των επίσημων ελέγχων, καλύπτονται από αυτές τις ε, μικροεπιχειρήσεις. Αποφασίσαμε πολιτικά κριτήρια. Θα πρέπει να υπάρξει αυτή η εξαίρεση να ξαναβάλουμε την υποχρέωση πληρωμής ε, στο κείμενο. Θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η ανεξαρτησία των ε, επιθεωρητών. με αυτά τα τέλη θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των ε, επιθεωρητών με μια εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κατάρτιση, καλύτερη κατάρτιση και θέλουμε να εξασφαλίσουμε επαρκή αριθμό. Είναι παράδεκτο να επισκεφτόμαστε μία φορά στα πέντε χρόνια ή μία φορά στα δέκα χρόνια τις επιχειρήσεις. Δεν λαμβάνουμε έτσι υπόψη τον κίνδυνο. Όχι, θα πρέπει να τις επισκεπτόμαστε με βάση μια ελάχιστη συχνότητα, την οποία βεβαίως θα καθορίσουμε συνεχεία. Και φυσικά η τα τέλη τα οποία συλλέγουμε δεν συλλέγονται για να πληρώνουν τον επιθεωρητή. Τα τέλη αυτά πηγαίνουν σε ένα κοινό κορβανά. Εδώ όμως ε, προσκρούμε στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Σε κάποια κράτη-μέλη, λόγω της εθνικής νομοθεσίας, το ποσό που εισπράτεται από τα τέλη ε, μπαίνει στον εθνικό κορβανά και θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να ξαναδώσει αυτά τα ποσά ε, για να φτιάξουμε ας πούμε σχολεία, αεροδρόμια, δρόμους. Με βάση άλλες εθνικές νομοθεσίες αυτά τα ποσά ξαναπηγαίνουν στις υπηρεσίες ελέγχου, απευθείας, διανόμου. Τώρα, πώς θα τα κάνουμε αυτά τα θέματα, ε, θα ευθυγραμμίσουμε, θα καθορίσουμε τα τέλη ανάλογα με τους φόρους που υπάρχουν σε εκείνο το κράτος μέλος, ε, δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε αυτό το κομμάτι. Σε κάποια κράτη-μέλη προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία ε, τα ποσά από τα τέλη να πηγαίνουν στο όλο σύστημα των ε, ελέγχων ε, για την διατήρηση αυτού του συστήματος. Τώρα, τα φυτά. Όλες οι τρίτες χώρες μπορούν να εξάγουν φυτά σήμερα σε εμά υπό τον όρο ότι σέβονται τους κανόνες. Υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο. Στα ζώα και στα, στο τομέα από πάντα το σύστημα είναι κλειστό. Η διεθνή, το Διεθνές Γραφείο Επιζωτιών το προβλέπει. Ενώ για τα φυτά υπάρχει πάντα, υπήρχε από πάντα ένα ανοιχτό σύστημα παρότι κάποιες τρίτες χώρες έχουν κλειστό σύστημα, το όλο παγκόσμιο σύστημα είναι ανοιχτό. Και εδώ πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση τελικά. Θέλουμε να έχουμε ένα κλειστό σύστημα όπως για τα, ζώα, όπως για τα προϊόντα ζωικής ε, προέλευσης, κάτι που δίνει κάποιες εγγύησεις βέβαια. Αυτό δεν αποκλεί βέβαια το να μπαίνουν ε, οι ε, έντομα επιβλαβείς οργανισμοί γιατί ξέρετε ότι συχνά ε, περίοδοι επόασης εδώ είναι πολύ πιο μεγάλες. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μία ασθένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μήνες ή χρόνο ή χρόνια μετά την εισαγωγή της. Ε, μια άλλη ερώτηση. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ασφάλεια ή στην ποιότητα. Η κυρία Οκόν Κον μιλησε για το πρόβλημα των ε, εμφυτευμάτων ε, μαστού που πιστοποιήθηκαν από εγκεκριμένους οργανισμούς ε, που είναι, ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα αλλά τις εποπτεύαν οι, διεθνείς, ε, οι δημόσιες αρχές. Συγγνώμη. Πρόκειται όχι για επίσημους οργανισμούς που κάνουν τους αρχικούς ελέγχους, αλλά πιστοποιημένους οργανισμούς που έχουν πιστοποιηθεί από τις εθνικές αρχές και κάνουν τους ελέγχους αυτούς. Αλλά στον τομέα της διατροφικής ασφάλειας ή στον τομέα της ποιότητας, δηλαδή ετικετοθεσία και τα λοιπά, ε, οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνε. Και θέλουμε οι εθνικές αρχές, οι επίσημες εθνικές αρχές, να συνεχίσουν να κάνουν αυτούς τους ελέγχους, με τη δυνατότητα όμως, εάν επιθυμούν, να εκχωρήσουν σε πιστοποιημένους οργανισμούς κάποιες αρμοδιότητες, αλλά που θα είναι πάντα υπό έλεγχο για να αποφύγουμε τέτοιους ελέγχους. Και στην περίπτωση των εμφυτευμάτων που μιλήσατε, ένας γερμανικό οργανισμό είχε επιστοποίησει ε, αυτά τα προϊόντα και από ό,τι φάνηκε ήταν αρκετά χαλαρό ο οργανισμό. Αν δεν ήταν το μέσο μου δεν μπορώ να μιλήσω για αυτόν. Πάντω, η δουλειά των ε, συναδέλφων μου επιθεωρητών από το γραφείο κτλ. και η δική μου είναι να επαληθεύουμε ότι εφαρμόζουν όλοι του ίδιου ελέγχου, ούτω ώστε το κράτο μέλο Α να μην είναι πιο χαλαρό από το κράτο μέλο Β που θα είναι πολύ πιο αυστηρό. Αυτά μπορώ να πω να μιλάω επί ώρε. Ναι κυρία Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι ο συναδελφός μου, ο Μάικλ, θέλει να προσθέσει κάποια πράγματα. Ναι. Ε, το ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ή θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένη να απαντήσει όλα. Θα σας παρακαλώ όμως να απαντάτε στις ερωτήσεις που σας έγιναν, όχι γενικά και αόριστα, επί παντός επιστητού, αλλιώς δεν θα προκάνουμε. Κύριο Σκάνελ. Σε σχέση με τα ερωτήματα που ε, μου αποτάνθηκαν και ως προς τις ε, περικοπές ε, των πόρων που διατίθενται μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας στον τομέα των τροφίμων ως προς την τροφική αλυσίδα και τους κτηνιατρικούς ελέγχους. Ε, μιλάμε λοιπόν για τις περικοπές. Εγώ θα πρέπει να ενημερώσω τον Γενικό μου Διευθυντή εάν υπάρχουν ε, μη αποδεκτοί κίνδυνοι που ανακύπτουν από την έλλειψη πόρων ή περικοπή πόρων έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο μας με τους υπάρχοντες πόρους. Ε, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα. Αλλά έχουμε κάνει οικονομίες Δηλαδή μειώσαμε την συχνότητα ελέγχων ε, στον τομέα της αλίας. Θα είχαμε περιοδικές, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε περιοδικούς ελέγχους σε πολλούς ε, εξαγωγείς, αλλά θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι έλεγχοι. Με βάση τη νέα πρόταση για τους επίσημους ελέγχους, Υπάρχει μια διάταξη όπου το Κοινοβούλιο θα έχει ε, πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα. Αν λοιπόν εγκριθεί αυτή η πρόταση θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε τι κάνουμε, ε, αν η συχνότητα είναι η αρμόζουσα και ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι πόροι, πόροι που διατίθενται δηλαδή έτσι ώστε να υπάρχει πιο στενός και αυστηρός η κυρία Μακέβων μίλησε για θέματα ποιότητας. Έθιξα εντάχει αυτό το θέμα των ποιοτικών ελέγχων. Όλοι οι έλεγχοι θα πρέπει να ε, βασίζονται σε μέρους ελέγχους που θα πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη. Δηλαδή πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια είναι η ιεράρχηση, δηλαδή εκεί που υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για την υγεία. Και πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ θεμάτων ασφάλειας ή ποιότητας, η ασφάλεια έχει προτεραιότητα. Γι' αυτό στις δικές μας επιθεωρήσεις βλέπουμε ότι στα πλαίσια των οργανικών γεωγραφικών δίκτων έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα από θέματα που άπτονται της ασφάλειας. Αυτό σχετίζεται και με τις απάτες. Όχι ότι δεν μας απασχολούν, αλλά η πραγματογνωμοσύνη αφορά θέματα ε, ασφάλειας. Ο μέσος κτηνίατρος δεν σημαίνει ότι ε, έχει την κατάλληλη κατάρτιση για να ασχοληθεί με θέματα καταπολεμιστής απάτης. Γι' αυτό χρειάζεται μια ευρύτερη πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι νέοι τομείς. Ευχαριστώ κύριε Χάρτμαν. Η κυρία Μακάβαν ρώτησε ε, πώς λειτουργεί το γερμανικό σύστημα ελέγχων και θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ αν έχετε ανταλλαγές με ομολόγους σας. Είμαι πολύ ικανοποιημένο με το γερμανικό σύστημα. Παντού βέβαια θα μπορούσε κάνει να έχει περισσότερο προσωπικό, αλλά όταν έχουμε ανταλλαγέ με συναδέλφους και άλλων ε, κρατών ε, μελών συνεργαζόμαστε πολύ καλά ε, και με την αμοιβαία κατάρτιση. Ποιο θα είναι ο μελλοντικό ρόλος των δημοσίων κτηνιάτρων και αν θα απορριθμιστεί. Το παράρτημα 2 δεν λέει τίποτα ε, για απορρίθμιση, αλλά το άρθρο 15 είναι πολύ ασαφές στη διατύπωση και ο φόβος μας είναι ότι η απορρίθμιση θα γίνει στη κατεξουδότηση πράξη από εκεί και πέρα, δηλαδή ότι θα χαρακτηρίζονται απαραίτητοι λιγότεροι έλεγχοι. Το δεύτερο, τι γίνεται με τους δημοσίους κτηνιάτρους ε, στην κρεοσκοπική ε, διαδικασία του ελέγχου. Σας είπα για το πακέτο γενής για την αλλαγή του κανονισμού 882. Οι κρεοσκοπικοί έλεγχοι ρυθμίζονται ε, ως, ε, ως αποσπασματικά και η ΕΦΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Τροφίμων, έχει πει αν να μην γίνονται εντομές στα σφάγια, λέει, να δεν ε, ε, βοηθάει για τον δημιουργισμό ορισμένων ε, ασθενειών και θα πρέπει να βελτιώνεται ο τρόπος με τον οποίο συνοδεύονται τα ζώα μέχρι το σφαγείο ή να γίνεται ανάντη και πάλι ο έλεγχος προηγουμένως. Υπάρχουν διάφορα σημεία που έχουν να κάνουν με το συνολικό πακέτο τα οποία έχουν εξαιρεθεί. Δεν ξέρω, ίσως στη συνέχεια πρέπει να ρυθμιστούν αυτά, αλλά τίθεται το ερώτημα αν είναι σωστή αυτή η αποσπασματική αντιμετώπιση. Πακέτο είναι δέσμη με το θέμα. Είναι το κόστος της, ε, του ελέγχου, όχι γενικότερα η κτηνοτροφία και η προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ κύριο Μπορέλο. Ε, δεν, δεν μου έχουν ε, αποτανθεί συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να στραφώ στη χρηματοδότηση των ε, μικροεπιχειρήσεων. Στην Ιταλία έχουμε απαλλάξει ε, τους μικρούς ε, λιανοπολίτες. Θεωρούμε όμως ότι ως προς επίσημους ελέγχους υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης σε αυτό το επίπεδο των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων της τάξης του 23%. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αναγκαίο ακόμα και εκείνη οι οποίοι ε, αποκλείονται από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αλλά συνεισφέρουν στον κίνδυνο αυτό, στον υγειονομικό ε, κίνδυνο, να πρέπει να συνεισφέρουν και χρηματικά. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε να συμπληρώσετε τίποτα κύριε Μπάνση, ε, δεν είστε υποχρεωμένος. Δεν μου έγιναν ειδικά ερωτήσεις σε μένα, Νομίζω ένα από τα σημεία που θέλω να τονίσω είναι η ανάγκη να βεβαιωθούμε ότι ό,τι καινούριο και να φέρουν οι προτάσεις να κρίνονται και να βασίζονται στο αποτέλεσμα. Ε, ε, σε ό,τι αφορά τις απάτες ή την εσκεμμένη μη συμμόρφωση δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί, να χτιστεί ένα ολόκληρο καινούριο σύστημα για να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει το σύστημα. Αυτό που θέλουμε είναι να αυξήσουμε την ασφάλεια και να γίνεται μια καλή ανταλλαγή ε, ενημέρωσης και πληροφοριών γρήγορα ε, και μέσω ενός συστήματος και μεταξύ των κρατών μελών. Σας παρακαλώ μην εφεύρουμε τίποτα καινούριο και άχρηστο και περιττό, αλλά να δημιουργήσουμε κάτι που θα μας βοηθήσει και να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία του και χρήση του στο πολύ σύντομο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Σεβάν δεν θέλει να απαντήσει. Η κυρία Λούλα Ιάντζη της έγινε να ρωτήσει πολλές. Το πρώτο ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχει απαλλαγή των μικροεπιχειρήσεων με βάση τη νέα καναδική νομοθεσία. Ναι, υπάρχει εξαίρεση, αλλά καθίσταται σαφές ότι η σημασία των μικροεπιχειρήσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ε, ε, βιομηχανία τροφίμων και ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία στην Ευρώπη από ό,τι στον Καναδά. Γι' αυτό θα επανέλθω ε, στον Καναδά επί του θέματος, γιατί δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο ε, λεπτομέρειας, ίσως καταγράφεται στους κανονισμούς, αλλά θα πρέπει να το ρωτήσω και μέσω γραμματείας θα σας ενημερώσω πώς έχει αυτός ο ορισμός των ε, μικροεπιχειρήσεων. Τώρα, ως προς την απάτη και το κυρωτικό πλαίσιο, η η νομοθεσία ε, στοχοθετεί θέματα ασφάλειας, αλλά και την πρόληψη στον τομέα της απάτης. Οι κυρώσεις μπορούν να φτάσουν στα 5 εκατομμύρια δολάρια και ως προς τις ε, ε, συλλογικές κυρώσεις μπορούμε να φτάσουμε από 250.000 σε 500.000 ανάλογα με την σοβαρότητα του αδικήματος. Αυτά τα στοιχεία ε, αναγράφονται στην ομοθεσία και για περαιτέρω ζητήματα θα σας δώσω τα στοιχεία που επιθυμείτε. Ναι, νομίζω θα αξιοποιήσει την ευκαιρία ο εισηγητής πολύ συγκεκριμένα να σας ρωτήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ε, όλους ε, που ήρθατε και μας μιλήσατε και απαντήσατε να περάσουμε αμέσως στο δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ. Χρειάστηκε και να περιμένετε πολύ. Τώρα είμαστε σε επιπτώσεις της πρότασης για τους επιχειρηματικούς παράγοντες και συνέπειες για τους καταναλωτές. Εισηγητής είναι ο κύριος Πυρίλο, ο οποίος θα αναλάβει την Προεδρία και θα διευθύνει και το πάνελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, ιδίως από την παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Πούντλε, από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, η πρόταση κανονισμού που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει κάποια καινοτόμα στοιχεία που έχουν σημαντική επίπτωση στους διάφορους οικονομικούς φορείς, επιχειρηματίες κτλ. του κλάδου. Η καινοτομία της πρότασης αφορά το γενικό τμήμα, τις επεκτάσεις, τις, τους υποχρεωτικούς επίσημους ελέγχους σε όλους τους τομείς της ε, διατροφικής αλυσίδας και την εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καθορίσει, να βασίσει τους ελέγχους σε, μια, σε ένα βάθρο που είναι κίνδυνοι. Κάτι άλλο που αφορά την τροποποίηση του 882 ε, είναι η χρηματοδότηση των ελέγχων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων διαφορετικό στοιχείο σε σχέση με τον 82. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Ντάβιντε Καλντερόνε που είναι ε, διευθυντής ε, του Κέντρου Διασύνδεσης του Μεταποιωτικών Βιομηχανιών Κρέατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εταιρείας Κιτράβη. Παρακαλώ, σας ευχαριστώ όλους. Καλησπέρα. Ε, είναι τιμή που βρίσκομαι εδώ να εκπροσωπήσω την, ε, τον κλάδο του ευρωπαϊκού κρέατος. Όπως είπε ο Πρόεδρος, ο τομέας του κρέατος είναι συνηθισμένος σε τέτοιες νομοθεσίες επί χρόνια τώρα. Στον κλάδο αυτό ε, υφιστάμεθα εκτινιατρικούς ελέγχους και υπάρχει και ένα καθεστώς ε, χρηματοδότησης, τελών δηλαδή. Το προβλέπει και 882 και αυτή η νέα πρόταση ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτό το στοιχείο, επεκτείνεται όμως αυτό το στοιχείο και σε άλλους τομείς. Ακούσαμε πολύ σημαντικές ερωτήσεις με το απόγευμα, ε, τι γίνεται με τις τρίτες χώρες, ε, ποια έμφαση δίνεται σε άλλους τομείς, σε άλλα προϊόντα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στον τομέα όμως, στον κόσμο του κρέατος, εμείς είμαστε συνηθισμένοι από την αρχή. Από πάντα είχαμε τέτοιου ελέγχου και εγώ θυμάμαι ότι όταν σφάζονται τα ζώα ε, η παρουσία των κτηνιάτρων πάντα ήταν υποχρεωτική. Επομένω, οι επιχειρηματίε ήταν απόλυτα συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο και επομένω δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υποβληθούν ε, σε αυτού του ελέγχου. Αυτό τώρα που για μα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και ο διευθυντή ο κ. Μπορέλο το τόνισε, είναι το θέμα του ανταγωνισμού. Δηλαδή, είμαστε σε μια κοινή αγορά, σε μια νέα αγορά, υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα θέλαμε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν την ίδια προσέγγιση για την εφαρμογή των ελέγχων και σε ό,τι αφορά τον αριθμό τους και σε ό,τι αφορά τη τιμή των ελέγχων αυτών και πώς χρηματοδοτούνται. Μας αρέσει η προσέγγιση Έλεγχο που βασίζεται στου κινδύνους, θα το δείτε και στην παρουσίασή μου, αλλά θα θέλαμε τα κριτήρια αυτού του, της θεωρητικής βαθμολόγησης των ε, επιχειρήσεων να, καθο, να καθορίζονται εκ των προτέρων, όχι από τα κράτη-μέλη, να αφήσουμε δηλαδή τις ε, αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αποφασίσουν ποιος αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο και να αποφασίσουν και τη συχνότητα των ε, τη συχνότητα των ελέγχων και εν συνεχεία τα τέλη. Τα τέλη τώρα, τα τέλη. Είναι σαφές ότι στον τομέα μας, σας είπα ότι επί, επί χρόνια είμαστε συνηθισμένοι να πληρώνουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πιστεύουμε ότι η διατροφική ασφάλεια και ότι η εγγύηση της ασφάλειας πέραν του ότι είναι ένα αγαθό και αφορά τη δημόσια υγεία, πέραν αυτού είναι σαφές ότι ο επιχειρηματίας ο οποίος παράγει κρέας ας πούμε είναι τμήμα, πολύ σημαντικό τμήμα αυτού του, αυτής εξίσωσης, αλλά όχι τα πάντα. Δεν αποτελεί τα πάντα. Επομένως, ε, η χρηματοδότηση των ελέγχων θα πρέπει να γίνεται και από την, α, τους φόρους του κράτους. Δεν είναι σωστό να πληρώνουμε απόλυτα εμείς για τους ελέγχους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποστούμε τους ελέγχους. Ε, συχνά η επίσημη έλεγχη είναι προσθέμενη αξία για την ε, επιχείρηση. Εγώ σας μιλάω για τις εξαγωγές από τρίτες χώρες. Ε, είναι αδύνατο να, γίνουν, να κάνουμε εμείς εξαγωγές σε τρίτες χώρες αν δεν υπήρχαν αυτοί οι επίσημοι έλεγχοι που μας δίνουν την ε, εγγύηση ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή. Αλλά είναι και μια σιγουριά και για τα καταναλωτή. Επομένως, ευπρόσδεκτη η έλεγχη, αλλά δεν είναι σωστό να πληρώνουμε τους ελέγχους 100% εμείς. Θα πρέπει να, ένα ποσό να, να πληρώνεται από τους φόρους του κράτους. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσέγγιση ότι ο έλεγχος βασίζεται στον κίνδυνο. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά πρέπει να δούμε, να διαφοροποιήσουμε από επιχείρηση σε επιχείρηση ποιε θα ελέγξουμε και πώς θα τις ελέγξουμε. Θα θέλαμε όπως τον κανονισμό να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία, επιπλέον στοιχεία, που αφορούν καταρχά τον, τον όγκο τη εμπορική δραστηριότητα, δραστηριότητας, την μην συμμόρφωση, αν έχει καταγραφεί μη συμμόρφωση στο παρελθόν, να υπάρχει δηλαδή ένα ρέκορντ, ας πούμε, ε, ένα αρχείο ε, για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θα, θα πρέπει να προβλέψουμε και αναδυόμενους κινδύνους, ε, παραδοσιακά στοιχεία. Σήμερα, με αυτές τις μέρες, συζητιέται κάτι πολύ έντονα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νέες μεθόδους επιθεώρησης για την παρουσία λογίσιου κρέατος στο Βόλιο. Πρόσφατα υποβλήθηκαν κατά της πράξη και τη ψήφισε του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αξιολόγηση των αναδυόμενων κινδύνων εντό αγωγικών έτσι, ε, οδήγησε την Κομισιόν, πολύ ορθά, στο να έχει μια διαφορετική προσέγγιση που να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Δηλαδή η επιθεώρηση των κρεάτων αν α πούμε δείξει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, από την υποθεώρηση και τον έλεγχο προκύψει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, να αλλάξουμε τη συχνότητα, να αλλάξουμε τον έλεγχο. Να έχουμε λοιπόν εστιασμένου ελέγχου που να βασίζονται στο πραγματικό κίνδυνο των προϊόντων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζει ο, μάλλον ο κανονισμός είναι η διαφάνεια. Εμεί ω επιχειρήσει δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δημοσιεύσουμε τα τα δεδομένα που έχουμε από του αυτοελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εδώ και πολλά χρόνια προβλέπει μία ευθύνη για την επιχείρηση ε, στον τομέα της ασφάλισης των τροφίμων. Η επίσημη ελέγχη είναι το ένα, η μία παράμετρος ευθύνη. Αλλά τελικά την τελική ευθύνη την έχει ο επιχειρηματίας. Κανένα πρόβλημα την αναλάβουμε σε αυτήν την ευθύνη. Ούτω ή άλλω τη λέει και, η δική μα νομοθεσία. Αλλά θα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα δεδομένα. Γιατί μιλάμε για διαφάνεια. Τι σημαίνει διαφάνεια, δεν πρέπει να κρύψουμε τα προβλήματα που μπορεί να έχουν στην επιχείρηση, αλλά πρέπει να τα διαχειριστούμε με σωστό τρόπο. Από τη συζήτηση που έγινε μέχρι στιγμή, προκύπτει συχνά το θέμα ότι ο επίσημο έλεγχος είναι μέσο για να αποκαλύψουμε απάτε στον τομέα αυτό. Εντάξει, προφανώ, Η απάτη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα στοιχείο. Αλλά κάποια στοιχεία μη συμμόρφωση και ξέρει πολύ καλά όποιο είναι επιθεωρητής γιατί μιλάω, Μερικέ αυτές, μερικές φορές αυτές οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δεν σημαίνουν ότι επίτηδες δεν συμμορφώθηκε η επιχείρηση. Κάνει, μπορεί να κάνει προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης, μπορεί να κάνει προσπάθεια ε, προσαρμογής στην νομοθεσία. Ε, οι παραγωγικές διαδικασίες να αλλάζουν, λαμβάνοντα ε, λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικές μελέτες κτλ. Δεν μπορεί να θεωρηθούν όλα αυτά μη συμμόρφωση, όλη αυτή η εξέλιξη και ο ε, επιθεωρητής μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιωθεί. Ε, η πρόταση του κανονισμού δίνει τη δυνατότητα σήμερα στους, ε, στους υπαλλήλους να δημοσιεύουν κάποια στοιχεία γενικά. Το θέμα είναι να έχουμε ε, λεπτομερή στοιχεία, μπορεί να είναι πολύ σημαντικά αυτά ε, και για την επιχείρηση και επηρεάζουν και τις, ε, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. δεν μπορούμε να τα δημοσιεύσουμε όλα γιατί υπάρχουν και θέματα εμπορικά, εμπορικά στοιχεία, εμπορικά μυστικά κτλ. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ε, να Ορίσουμε πολύ καλά τις έννοιες απάντη, απάτη και μη συμμόρφωση. Το θέμα της χρηματοδότησης, πάρα πολύ σημαντικό. Το είδαμε ότι με τη σημερινή πρόταση προβλέπουμε δύο είδη χρηματοδότησης, άμεση χρηματοδότησης. Δύο κριτήρια που υιοθετούμε. Στη μία περίπτωση μιλάμε για το κόστος της επιθεώρησης, πόσο κοστίζει δηλαδή ο έλεγχος, και στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για τέλη τα οποία θα καθοριστούν ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ελέγχεται ή όχι η επιχείρηση. Και στις δύο περιπτώσεις εμείς θα θέλαμε να προβλεφτεί η δυνατότητα όχι μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό ελέγχου, δεν μας φοβίζει αυτό. Να πληρώνουμε λιγότερα όμως σε περίπτωση ε, που έχουμε να κάνουμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ε, σωστές ας πούμε. Αν δηλαδή μια επιχείρηση όταν ελέγχεται είναι πάντα ακριβή, ε, συμμορφούται κτλ. Θα θέλαμε τη δυνατότητα να έχει μια έκπτωση, να πληρώνει λιγότερα τέλη. Αυτό δεν ισχύει όμω. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο και νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίση άλλο σημαντικό στοιχείο είναι, και εδώ επανέρχομαι σε κάτι που υπόθηκε ήδη πριν, είναι σημαντικό η έλεγχη και αυτοέλεγχη που κάνει η επιχείρηση, που είναι τόσο πολύ, να λαμβάνονται υπόψη. Γιατί ο αυτοέλεγχο όχι μόνο αυτοχρηματοδοτείται, χρηματοδοτεί δηλαδή την επιχείρηση, αλλά οι αυτοέλεγχοι συνδέονται και με άλλα ε, θέματα. Έχουμε του επίσημου ελέγχου ε, που συνδέονται με τα κτηνιατρικά θέματα και του αυτοελέγχου που συνδέονται με τα εμπορικά θέματα. Ε, οι επιχειρήσει ε, πρέπει να κάνουν μια σειρά από ελέγχου, από αναλύσεις, πολύ συγκεκριμένε κτλ. Γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη μα καθόλου αυτέ τις στιγμέ αυτά τα στοιχεία, κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων. Ειδικά όταν η έλεγχη και η αυτοέλεγχη έχουν ακριβώ τον ίδιο στόχο κάποιε φορέ. Είναι πολύ σημαντικό επίση αυτό. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για να μειώσουμε το κόστο του ελέγχου είναι αυτό που ρωτάμε εμεί. Ειδικά στον τομέα του κρέατο, κάποιε δραστηριότητε του επίσημου ελέγχου, όπω προβλέπει ήδη νομοθεσία, ειδικά στον τομέα τη φαγή, από προσωπικό το τεχνικό που έχει υποστεί κατάρτιση που δεν είναι κατά ανάγκη κτηνίατρος με πανεπιστημιακό δίπλωμα και που πρέπει να τον πληρώνω και περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον δόκτωρα Καλντερόνε. Ακούσαμε την ε, άποψη από το τομέα του κρέατος. Τώρα περνάμε σε έναν άλλο τομέα, εξίσου σημαντικό, που αφορά τους σπόρους όπου η Ευρώπη είναι ο πρώτος παγκοσμίος παραγωγός όπου θα πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των καλλιεργειών, δηλαδή τα οποροκυπευτικά τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι μας. Δίνω το λόγο στον κύριο Μάσιμο Μπιλόνι, που είναι Γενικός Διευθυντής του τομέα ε, διαχείρισης των σπόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ του τομέα των σπόρων και να μιλήσω για τη συνεισφορά των σπόρων στην διατροφική ασφάλεια και πώς οι επίσημοι έλεγχοι ε, δρούν θα μιλήσω εξ ονόματος της European Seed Association, αλλά θα σας μιλήσω και για συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Θα σας μιλήσω για τη δική μας ε, Ιταλική επιχείρηση που εμπίπτει στις ΜΜΕ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους επίσημους ελέγχους και πώς έμπρακτα ε, έχουν επιπτώσεις. Προσπαθώ να σας δείξω πως έχει ο τομέας των σπόρων. Αφορά ε, περίπου 7.000 επιχειρήσεις. Ε, το 70% ε, εμπίπτουν στον τομέα των μικροεπιχειρήσεων. Μιλάμε για 7 δις ευρώ τζίρο. Συμμετέχουν 50.000 εργαζόμενοι, ένα τέταρτο των οποίων οποίων ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη. Οι, επενδύουν το 20% του τζίρου αυτές οι επιχειρήσεις του κύκλου εργασιών σε νέες επενδύσεις, κάτι το οποίο μας κάνει τον υπαριθμόν ένα παραγωγό ε, παγκοσμίου στον τομέα των σπόρων. Ε, σε σχέση με τους πόρους ε, θα σας μιλήσω εντάχει ε, από ένα κιλό σπόρων μπορούμε να φτάσουμε σε 500 κιλά και αυτό αφορά και τον τομέα των, της ντομάτας που μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ μεγάλο τζίρο Μπορούμε να έχουμε λοιπόν ευρύτατη προστιθέμενη αξία, αλλά αν δεν γίνει σωστός έλεγχος και διαχείριση, τότε θα έχουμε περισσότερες ασθένειες και παρουσία παρασίτων, καθώς και προβλήματα ποιότητας καθαρά. Για να σας μιλήσω για τη δική μου επιχείρηση, είναι μια επιχείρηση που ε, παράγει στο Βερτσέλι στη Βόρεια Ιταλία ε, σπόρους ρυζιού. Πρόκειται για 13 ε, εκμεταλλευτές και δεν πρέπει να ξεχνάμε το Πιεμόντε και η Σαρδινία είναι επικεφαλής αυτής της παραγωγής. Υπάρχει και ένα ερευνητικό κέντρο και τρεις μονάδες επιλογής. Έχουμε λοιπόν παραγωγή σπόρων που διατίθενται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και μιλάμε και για μία ε, πιστοποίηση και θέση εμπορία σε όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη. Έχουμε ένα κύκλο εργασιών 9 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή είμαστε πάνω από τις μικροεπιχειρήσεις. Έχουμε 12 εργαζόμενους, άρα εμπίπτουμε όχι στις μικροεπιχειρήσεις αλλά πολύ κοντά σε αυτές. Εμείς ως ΜΜΕ στο τομέα της παραγωγής σπόρων θέλουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα, ποιοτική παραγωγή μέσα στα πλαίσια της τροφικής αλυσίδας. Σας μιλώ για την παραγωγή ριζότο στην, στην Ιταλία, παέλια στην Ισπανία και ούτω καθεξής. Μιλάμε για πιστοποιημένες ποικιλίε δηλαδή σπόρων. Ως προς τους ελέγχους στον τομέα των σπόρων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανέκαθεν υπήρχαν έλεγχοι στον τομέα των ε, σπόρων εδώ και 40 χρόνια και οι έλεγχοι αυτοί είχαν σαν στόχο τα ποιοτικά προϊόντα, τα οποία να είναι υγιή προϊόντα, υγιεινά προϊόντα, μέσα στα πλαίσια μία συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Όταν μιλάμε για ελέγχους, ε, τι εννοούμε. Στον τομέα των σπόρων υπάρχει αρχικά ένας έλεγχος in situ, εκεί δηλαδή που ο αγρότης παράγει, καλλιεργεί, για να μιλήσουμε για την ταυτότητα των ε, ποικιλιών και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν ασθένειες πριν φτάσουμε στην ε, σπορά. Ε, μιλάμε λοιπόν για σπόρους που δεν είναι για ανθρώπινη κατανάλωση ακόμα. Γίνεται αποθήκευση και εκεί λαμβάνονται δείγματα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν παθογόνοι παράγοντες ιδιαίτερα ε, έτσι ώστε να μιλάμε για να μην υπάρχουν παθογένειες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι και αλλιώς στην επικράτειά μας. Μετά τη συσκευασία γίνονται επίσης έλεγχοι πριν να τεθεί σε, στο εμπόριο το προϊόν και μετά μπαίνει στο εμπόριο το, ο σπόρος, διαφορετικά αποκλείεται από το εμπόριο. Έτσι, ο τομέας αυτός ε, διέπεται από μία ανιχνευσιμότητα, πλήρη ανιχνευσιμότητα και έτσι οι αγρότες που προβαίνουν σε αυτές τις ε, σπορές έχουν να κάνουν με ένα προϊόν ε, το οποίο πραγματικά είναι υγιεινό. Για τους ελέγχους ε, καταβάλουμε 450.000 ε, ευρώ, δηλαδή το 5% του κύκλου εργασιών μας. Ποιοι είναι οι στόχοι των επίσημων ελέγχων, γιατί θεωρούμε ότι είναι χρήσιμοι επίσημοι έλεγχοι. γιατί όλη η, παραγωγή, όλη η αλυσίδα παραγωγής ή καλλιέργειας είναι ισότιμη και εγγυάται και η προστασία, η προστασία των καταναλωτών. Δηλαδή μιλάμε για ένα σαφώς αναγνωρίσιμο προϊόν αυτός ο σπόρος που καλλιεργείται δηλαδή από το γεωργό για να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο αγαθό για το που προέρχεται για το εμπόριο να ξέρουμε από πού προέρχεται. Επίσης ε, με τον έλεγχο του σπόρου δεν έχουμε τη διάδοση ασθενειών και παθογόνων παραγόντων που αφορούν ε, παθογένειες που θα έπρεπε να μπουν σε καραντίνα. Διαφορετικά ε, δεν θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε τη διάδοση ορισμένων ασθενειών. Τι σκεφτόμαστε για το μέλλον. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος, ε, μεγαλύτερη εναρμόνιση και ολοκλήρωση των επισήμων ελέγχων στον αρμόδιο φορέα και επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο που να διέπει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά αυτό επιχειρήσεις όπως η δική μου που εντάσσεται στις ΜΜΕ και που θέτει το προϊόν της στο εμπόριο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τη δραστηριότητα της δικής μας ΜΜΕ που εξάγει σπόρους ρυζιού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για 1,5 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ο κύκλος εργασιών μας και μιλάμε και για ένα κύκλο εργασιών της τάξης του 5% εκτός Ευρώπης, της 5% σε σχέση με τη συνολική μας, το συνολικό μας τζίρο. Θα πρέπει όμως να υπάρξει μία πλούστευση του πεδίου δραστηριότητας, να μην υπάρχει ένα υπερβολικό κόστος λειτουργίας και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν επίσημοι έλεγχοι από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σπόρων. Θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και τα σε επανδρομένα εργαστήρια, έτσι ώστε παράλληλα με την επίσημη δραστηριότητα να υπάρχουν και έλεγχοι Δηλαδή πριν από την καλλιέργεια ή παραγωγή του σπόρου να ξέρουμε αν η ποιότητα είναι καλή. Για να μην έχουμε ε, παρτίδες οι οποίες απομακρύνονται από την αγορά. Άρα αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να επισημοποιηθεί έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα του προϊόντος με δειγματοληπτικούς ε, ελέγχους επιθεώρησης. Αυτό είναι ζωτική σημασία για τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, μπορούν να έχουν μια πιστοποίηση και μια επιθεώρηση χωρίς υπερβολικό κόστος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι ΜΜΕ στον τομέα των σπόρων αφορούν το 70% απορροφούν το 70% της δραστηριότητας, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει επιπρόσθετο ε, κόστος ε, ελέγχων. Για να επιταχύνω θα ήθελα να πω ότι ως προς την ανιχνευσιμότητα θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες ε, προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται στον τομέα αυτής της βιομηχανίας σπόρων και ελάχιστες προδιαγραφές εναρμόνισης. Στη περίπτωση του ρυζιού που είναι ένας βασικός τομέας θα πρέπει να γίνει συσκευασία με την ονομασία της ποικιλία. Άρα ξεκινάμε από έναν επίσημο έλεγχο και μόνο έτσι μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι αναφέρεται αυτή η συγκεκριμένη ε, ποικιλία. Τώρα, ως προς τα συμπεράσματα θεωρώ ότι ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σπόρων θα πρέπει να υπάρχει το επίσημο ε, σύστημα ελέγχων και να γίνει εναρμόνιση αυτού του συστήματος σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη για να υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβαση στην αγορά καθώς και συνέργεια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να εγγυηθούμε την ποιότητα και την ανιχνευσιμότητα του τομέα αυτού που ξεκινάει από έναν απλό σπόρο. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρα Μπιλόνι. Ακούσαμε διάφορα στοιχεία για τους ελέγχους, ε, ούτως ώστε να έχουμε ελεγχόμενους σπόρους, οι οποίοι μετά μπαίνουν στην αγορά και ακούσαμε ότι οι σπόροι Έχω μια υψηλή προστιθεμένη αξία. Εξού και η σημασία τους. Θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση του κυρίου Λουκ Πέτερς, πρόεδρος της ομάδας εργασίας Κόπα Κοζέκα για τα φυτο ζητήματα. Ε, είναι μία από τις πιο σημαντικές, σημαντικούς συνεταιρισμούς. Ξέρω ότι με την παρουσίασή του θα μας μιλήσει για την επίπτωση της πρότασης για τους τρόπους, σε ό,τι αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των ελέγχων. Ιδίω επιπτώσεις που θα έχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικροεπιχειρήσεις. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που ε, προσκαλέσατε και την κόπα Κοζέκα που εκπροσωπεί ε, τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, πολλά από τα μέλη μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εντάσσονται στην πρόταση ως προς το ε, χρηματοδοτικό σκέλος και τι σημαίνει αυτό για τους μικρομεσαίους. Από πλευράς Κόπα Κοζέκα θα θέλαμε να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των το ανεξάρτητο των ελέγχων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς. Αυτό έχει να κάνει και με την καθημερινή μας ενασχόληση με την παροχή τροφίμων ε, και μάλιστα ασφαλών και υγιεινών. Οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι συνεταιρισμοί είναι θύματα όλο και αυξανόμενου ανταγωνισμού, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εξωτερικούς ε, παγκόσμιους και καλούνται να ε, ανταποκριθούν σε πολύ ψηλές προδιαγραφές. Ο σωστός και υγιής ανταγωνισμός βοηθάει και για την καινοτομία και για την ασφάλεια των τροφίμων, για το κλίμα, για το περιβάλλον, για μια σειρά θεμάτων και για την αντιμετώπιση των νέων αδειωμένων κινδύνων. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός λειτουργεί σωστά όταν εντάσσεται σε ένα ε, περιβάλλον ίσων κανόνων παιχνιδιού για όλους τους φορείς και τους ενεχομένους συμπεριλαμβανομένων και κρατών. Ε, είναι πέρα από την εσωτερική αγορά αυτά και ως αγρότες εμείς λυπούμεθα που η παρούσα αναθεώρηση δεν έχει λάβει παντού υπόψη της αυτό το θέμα. Ε, μερικοί από τους βασικούς εταίρους μας έχουν ακόμα κρατικές ενισχύσεις και επίσης πολλές φορές οι Ευρωπαίοι φορείς ε, και εταιρείε θα πρέπει να πληρώνουν τις περαιτέρω ελέγχους ε, που επιβάλλουν οι τρίτες χώρες όταν εξάγουμε τα προϊόντα μας. Δηλαδή βάζουμε δύο φορές το χέρι στην τσέπη. Παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνουμε στη χώρα μας ή στην περιφέρεια μας και μετά πρέπει να πληρώνουμε και τον πελάτη για να κάνει έλεγχο στη χώρα προορισμού. δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το κόστος αποκλειστικά τους ιδιώτες ανεξαρτήτως μεγέθους. Από ότι η φύση του αυτό ε, είναι κατά του ανταγωνισμού. Η επίσημη ε, ελεγχή θα πρέπει να θεωρείται δημόσια κοινοφελής υπηρεσία, την οποία ήδη έχουμε χρηματοδοτήσει από το φορολογικό μας σύστημα. Γι' αυτό το λόγο απορρίπτουμε ένα υποχρεωτικό σύστημα τελών ανεξαρτήτως ε, μεγέθους της επιχείρησης. Δεν ακούστηκε αυτό προηγουμένως, αλλά πολλά νοσήματα ε, και των φυτών και των ζώων ε, έρχονται μέσω του τουρισμού και των ταξιδιωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ακούστηκε ακόμα σήμερα. Και αυτοί πώς συνεισφέρουν στο σύστημα ελέγχου οι άνθρωποι. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαιρούνται από το κόστος ε, των επίσημων ελέγχων. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί. Σήμερα ισχύει. Θα πρέπει όμως να να, μην επιβαρύνονται όλες οι επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες εκπροσωπούν ε, την καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και εξαίρεσή τους ε, εγγράφεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής για το 2020 και την ελεγχιστοποίηση του γραφειοκρατικού άχθους ε, για τις μικρομεσαίες έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με τη Eurostat στις μεγάλες επιχειρήσεις η συμμετοχή τους ε, είναι πολύ μικρή σχετικά με τον τζίρο τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρομεσαίες είναι μόνο 5% του συνολικού τζίρου των κλάδων αυτών. Συμφωνώ ότι είναι πολλές οι μικρομεσαίες που συμμετέχουν. Αν δείτε όμως τον κύκλο εργασιών είναι μόλις 5%. 95% λοιπόν οι 90% μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτουν μόλις το 5% του τζίρου. Επίσης δεν υπάρχει ισορροπία την εξουσία της τροφικής αλυσίδας ε, και δεν μπορούν αυτές πλέον οι εταιρείε να μετακυλήσουν το κόστος στον καταναλωτή. Ήδη αυξάνεται το κόστος των ε, ε, γεωργικών εφοδίων έτσι κι αλλιώς και έχουμε πολύ μεγάλη επιφάνηση για να πληρώνουμε και το κόστος των επιθεωρητών ε, σε επίπεδο εκτροφής. Ενώ η εκτροφή δεν μπορεί να συμπιέσει το κόστος ούτε να το μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή στην τροφική αλυσίδα που είναι μερικούς κρίκους πιο κάτω από την εκτροφή. Θα πρέπει το κόστος να το επομίζονται και άλλοι φορείς και οι αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε σχέση με όλα αυτά. Δυστυχώς δεν έχουν δοθεί και κίνητρα ούτε σαφείς προϋποθέσεις από τις αρμόδιες αρχές για να γίνονται οι επίσημοι έλεγχοι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τι σημαίνει αυτό. Ότι στον πραγματικό κόσμο τελικά την ύφθα την πληρώνει πάντα ο παραγωγό. Αυτό είναι παράδεκτο. Εντάξει, είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε υγιεινή τρόφιμα. Δεν αμφιβάλλουμε και δεν το αμφισβητούμε. Συμφωνούμε απολύτω. Αλλά δεν θα πρέπει μόνο εκείνοι που παράγουν τρόφιμα να επομίζονται το 100% του κόστου των ελέγχων. Και φοβούμαστε πάρα πολύ. Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εντάξει οι μεγάλοι αριθμοί που ακούστηκαν, αν πρέπει να επιβαρυνθούν με ένα νέο φορολογικό σύστημα θα φαγωθούν όλα τα λεφτά στη λειτουργία του συστήματος ελέγχων τελικά. Να σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι συμβαίνει σήμερα στις εκτροπές μας. Οι γεωργοί και αγρότες ήδη έχουν αυξημένους ελέγχους σε διάφορα χρονικά διαστήματα που ε, είναι και χρονοβόρες και ε, χρήματα ε, κοστίζουν θα πρέπει να ενοποιούνται οι έλεγχοι και να ομαδοποιούνται κάπως. Πολύ συχνά οι αγρότες ε, συμμετέχουν σε θελοντικά συστήματα ελέγχου που ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μερικές φορές ξεπερνούν κιόλας. Αυτά τα εθελοντικά συστήματα έχουν και επιχειρήσεις και ελέγχους από ανεξαρτήτους και πολλές φορές πιστοποιημένους φορείς και ελέγχουν όλες τις νομικές απαιτήσεις ε, και τις υποχρεωτικές αλλά και τις προαιρετικές. Τι συμβαίνει λοιπόν στην πραγματική ζωή. Κάνουμε αυτό τον έλεγχο και την άλλη μέρα έρχεται ο επίσημος έλεγχος. Χαίρετε, ήρθαμε να σας ελέγξουμε. Το πληρώνουμε και εμείς πάλι και ε, ελέγχουμε ακριβώς τις ίδιες δραστηριότητες που προηγουμένως είχαμε ελέγξει. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ιδιωτικοί έλεγχοι και επίσημοι δημόσιοι θα πρέπει να μπορούν να συνενωθούν να συνδυαστούν και πάλι θα γίνουν εκεί μεγάλες οικονομίες από αυτή τη συνέργεια και θα είναι και πιο αποτελεσματικός και πιο συντονισμένος ο έλεγχος. Όχι μόνο μεταξύ των αρμοδίων αρχών αλλά και με, με ε, επίσημα πιστοποιημένα ε, μέρη που κάνουν τους ελέγχους. Και καλωσορίζουμε βεβαίως πάντα τη διαφάνεια και την εναρμόνιση όπως αυτή προτείνεται και για τις αρχές και για τους φορείς ε, του κλάδου. Και βέβαια θέλουμε καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ε, καλές πρακτικές για την αποτελεσματικότητα να διαβιβάζονται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα πρέπει να έχουμε όμως κανόνες που να εγγυώνται την ανταγωνιστικότητα ε, των γεωργών μας και των συνεταιρισμών μας με έναν τρόπο πιο ευφύ για τη χρήση των υφισταμένων πόρων ενώ πάντα θα διατηρούμε την υψηλή ποιότητα παραγωγής και προδιαγραφών. Η Ευρωπαϊκή ε, παραγωγή και οι Ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί θέλουν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το έχουν αυτό υπόψη τους και να δώσουν εκεί την έμφαση στην αναθεώρηση της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον δόκτωρα Πέτερς, ο οποίος μας εξέθεσε τη σκέψη του που είναι άκρος ενδιαφέρουσα και θα αξιοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης. Δίνω το λόγο στην ε, δόκτωρα Ρουθ Βεάλε που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΕΜΒΗ που μας προσκάλεσε για να παρουσιάσουμε κάποια από τα βασικά θέματα ε, και τη σκοπιά των καταναλωτών. Πολλά από τα θέματα ε, βλέπω ότι έχουν συμπεριληφθεί σε κάποια άλλη παρουσίαση. Αλλά μίλησε κυρίως ε, για τους επίσημους ελέγχους. Εκείνη θα ήθελα να σταθώ πολύ σύντομα, να διατάξω πολύ σύντομα αυτό το θέμα σήμερα. Πρώτο θέμα είναι αυτό. Αν θέλουμε να χτίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ε, διατροφική αλυσίδα, είναι σημαντικό αυτό. Ε, ακούσαμε διάφορους τομείς όπου η εμπιστοσύνη των καταναλωτών διαβρώθηκε τα τελευταία χρόνια και αν θέλουμε πραγματικά οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη, ε, είναι σημαντικό η επίσημη έλεγχοι ή να γίνονται ανεξάρτητα ε, από τις αρμόδιες αρχές. Και οποιοδήποτε φορείς συμμετέχουν είναι Είναι σημαντικό να έχουμε τακτικούς ελέγχους, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι φορείς αυτοί ασκούν τα καθηκόντά τους πολύ σωστά. Το θέμα δεν είναι ποιο κάνει του ελέγχου τη αλλά γιατί πρέπει να καλύπτουν αυτέ οι επιθεωρήσει και ποιο πρέπει να ελέγχεται. Ε, εδώ προκύπτει πάλι το σκάνδαλο του αλογισιού κρέατος. Είναι το πιο πρόσφατο μεγάλο σκάνδαλο στην Ευρώπη και τονίζει ότι όλοι οι ενδιάμεσοι ε, πρέπει να καταχωρούνται για νομικούς λόγους. Είναι σημαντικό αυτό. Ε, το σκάνδαλο αυτό έδειξε ακόμα μια φορά πόσο μακρά και περίπλοκη είναι αυτή η διατροφική αλυσίδα και πρέπει να πραγματικά να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι ενδιάμεσοι υπόκεινται σε κάποιες νομικές υποχρεώσεις. Φυσικά θα πρέπει οι πόροι να, επειδή είναι συγκεκριμένοι, ε, να εστιάζουμε στις επιχειρήσεις και στις δραστηριότητες που είναι πιο επικίνδυνες. Όταν μιλάμε για επικίνδυνες, για κίνδυνο, το είπαν και πολλοί ευρωβουλευτές, θα πρέπει ο κίνδυνος να συμπεριλαμβάνει και το, την οικονομική απώλεια των καταναλωτών και τον κίνδυνο του να σε παραπλανήσουν πέρα από το, τη ζημιά στην υγεία. Από τις πρόσφατες κρίσεις είδαμε ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ποιοτική τροφή, ποιοτικά τρόφιμα και ότι πληρούν τα πρότυπα ε, ασφάλισης των τροφίμων, όλα τα προϊόντα αυτά, τα διατροφικά που κυκλοφορούν. Επίσης, από τα πρόσφατα σκάνδαλα πάλι προκύπτει σημασία ε, στενού συντονισμού, επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, όπω είπε και ο εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να είναι, υπάρχει ένα στέρεο και αποτελεσματικό σύστημα που επιτρέπει γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το είπε και η Κομισιόν και προβλέπεται από την πρότασή τη. Γρήγορη διασπορά των πληροφοριών για πιθανού κινδύνου. Αυτό ε, ίσως ε, είναι το αποτελεσματικό ε, στοιχείο για να σταματήσουμε το πρόβλημα στην πηγή. Ε, μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι ρηπογόνε ουσίε και να τι σταματήσουμε κοντά στην πηγή. Είναι σημαντικό να υπάρχει το δίκτυο επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, μια πιθανή απειλή κτλ. Ε, να αρχίσουν οι τροχοί να κινούνται, ούτω ώστε οι καταναλωτέ να ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν, ούτω ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητε δράσει. Όλοι οι μιλητέ μίλησαν για την χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων. Τεράστιο θέμα αυτό. Ε, Προφανώ το επόμενο μήνε θα συζητήσει πολύ το Κοινοβούλιο αυτό το θέμα. Φυσικά όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν επαρκεί πόροι για την εφαρμογή τη νομοθεσία για τα τρόφιμα. Η Κομισιόν προτείνει να επεκτείνει τη συλλογή των τελών σε μια ευρύτερη αλυσίδα επιχειρήσεων. Υπάρχει επίσης η εστίαση στη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των τελών και την ίσπραξη των μελών. Είναι σημαντικό αυτό, να είναι η όλη διαδικασία ώστε να τον πιο διαφανή, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχέ ε, είναι σίγουρα ανεξάρτητε, δεν αμφισβητείται η ανεξαρτησία τους ή δεν θεωρείται ότι δεν είναι ανεξάρτητε. Επίσης, ε, μπορεί τα τέλη να εισαχθούν τόσο ώστε να δοθούν ε, κίνητρα στη βιομηχανία στον κλάδο για να συμπεριφέρεται σωστά. Ε, όπως είπε και ο Ιταλός ε, εκπρόσωπος, οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με, το, με τον νόμο μπορούν να υποφεληθούν από μείωση των τελών. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και το αντίστροφο. Εάν συνέχεια παραβαίνει, θα πρέπει να αυξάνονται τα ποσά που πληρώνεις, τα τέλη που πρέπει να πληρώσεις. Ένα ερώτημα ερωτηματικό που έχουμε και νομίζω ότι ακούστηκε από πολλούς άλλους σήμερα. Είναι η εξαιρέση για τις μικροεπιχειρήσεις. Μιλήσαμε για μια προσέξη να βασίζεται στον κίνδυνο στις επιθεωρήσεις και στον τρόπο διενεργειάς τους. Και ξέρω ότι οι μικροεπιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, γιατί μπορεί και αυτές να αποτελούν κίνδυνο και υψηλό κίνδυνο. Γιατί θα πρέπει ε, να έχουμε μία προσέγγιση με στον κίνδυνο για τους επίσημους ελέγχους, αλλά όχι για τον υπολογισμό των τελών. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να το συζητήσει νομίζω η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επανερχόμαστε στο θέμα φυσικά των προειδοποίητων ελέγχων, των ευθύντων ελέγχων. Αυτό για μας είναι τεράστια σημασία. Πρώτερη προειδοποίηση θα πρέπει να δίδεται μόνο σε εξαιρετικέ περιπτώσεις. Και με στην πρόταση της Κομισιόν ε, Υπάρχει ένα ερωτηματικό για το ποιες είναι αυτές οι συνθήκες ε, υπό τις οποίες προαναγγέλλονται οι έλεγχοι. Για μας, αν προαναγγείλεις μια επιθεώρηση, έστω και λίγες ώρες πριν, ο υπεύθυνο ε, ε, που θα πάει εκεί μπορεί να μην καταλάβει ποια είναι η συνήθιση πρακτική της επιχείρησης. πρέπει να, διευκρινιστούν το ποιες αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις υπό τις οποίες δεν προαναγγέλλεται, συγγνώμη, υπό τις οποίες μάλλον προαναγγέλλεται ο έλεγχος. Θα πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα να των απροειδοποιητών ελέγχων. Το θέμα των κυρώσεων επίσης ακούστηκε πολλές φορές. Ο Επίτροπος επίσης το είπε ότι οι παραβάτες πρέπει να πληρώνουν και όλοι το πιστεύουμε εδώ. Προφανώς υπάρχει ανάγκη για τσουχτερά ε, πρόστιμα. Φυσικά αυτό είναι ένα αντικίνητρο για παραπλανητικές, μη ασφαλείς πρακτικές, για απάτες κτλ. Το θέμα προσυζήτηση είναι φυσικά για το πώς λειτουργεί το όλο θέμα αυτό στην πραγματικότητα. Θα θέλαμε να διερευνήσουμε λιγάκι το ρόλο της Κομισιόν για να αναπτύξει κατευθυντήρες γραμμές ε, για τα κράτη-μέλη. Γιατί όπως ακούσαμε η νομοθεσία, οι νόμοι λοιπά εφαρμόζονται διαφορετικά. Επομένω, αν υπάρχουν κατευθυντήρε γραμμέ, βοηθηθούν τα κρατη για να εφαρμόζουν με συνεπή τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, το θέμα των κυρώσεων. Και το θέμα της διαφάνειας της συμμόρφωσης είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα υπόλοιπα στον κατάλογο, αν υπάρχουν και δεν υπάρχει διαφάνεια για τη συμμόρφωση, τότε οι καταναλωτέ δεν θα ξέρουν και δεν θα έχουν την εμπιστοσύνη στην αλυσίδα αυτή, τη διατροφική. Υποστηρίζω τον εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε το σύστημα που έχουν εκεί, της τηλίτευσης. Δεν υπάρχει μόνο εκεί, αλλά και στη Δανία και σε άλλα κράτη-μέλη, όπου συζητούν τη δυνατότητα εισαγωγή του. Και από αυτά που ξέρουμε από τρίτε χώρε όπου αντίστοιχα συστήματα έχουν εφαρμοστεί, είδαμε ότι έχουμε μείωση σε τροφικές δηλητηριάσεις ε, σε αυτά τα κράτη-μέλη που ένα τέτοιο σύστημα. Είναι σημαντικό οι καταναλωτές να έχουν πληροφορίες για τα πρότυπα ε, και το επίπεδο συμμόρφωσης όλους τους, όλων των φορέων της αλυσίδας, όλων των εμπλεκομένων και αυτό θα είναι επωφελές καταρχάς για τους καταναλωτές. Μπορείς να επιλέξεις με τα λόγω γνώσεως τι Πού θες να αγοράσεις, τι θες να αγοράσεις, τι θες να φας. Και κατά δεύτερον, όπως προαναφέρθηκε, θα μας βοηθήσει κάτι τέτοιο να έχουμε ακόμα πιο υψηλά πρότυπα. Άρα θα είναι πολλά τα ωφέλη. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των ελέγχων τους και υπάρχουν όμως και επιχειρήσεις που θα πρέπει να, είναι, να υποχρεώνονται να δημοσιοποιούν αυτά τα στοιχεία και να δίνουν αυτές τις πληροφορίες στους καταναλωτές ούτω ώστε ο καταναλωτή, όπω είπα, να αποφασίζει ξέροντα τι αποφασίζει. Μετά από τη σημερινή συζήτηση, ε, νομίζω ότι έχετε πολλά που μπορείτε να σκεφτείτε. Περιμένουμε τη συνεργασία μαζί σας τους επόμενους μήνες. Να, θέλουμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Δυστυχώς θα πρέπει να φύγω, δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, αλλά φυσικά αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή με εμάς. Ευχαριστούμε. Ναι, να δώσω το λόγο στον ε, πρόεδρο Κλάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συμμετέχοντες και την κυρία η οποία εξέφρασε την άποψη των ε, καταναλωτών ε, με στα πλαίσια των διασφαλίσεων από τους ελέγχους των προϊόντων, ιδιαίτερα εντός Ευρώπης. Έχετε το λόγο για να ανοίξει η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πυρή. Είχαν την καλοσύνη ε, και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι από την άλλη πλευρά του κλάδου να μας δώσουν τα επιχειρήματά τους και καλό είναι έτσι, ακούμε όλες τις πλευρές γιατί έχουμε ένα κοινό στόχο και κοινό δρόμο προς τα εκεί. Θα παρακαλέσω τους κοιόδης συζητητές να μας πούν αν έχουν ερωτήσεις ή τους λοιπούς συναδέλφους. Ο κύριος Σνέλχαρτ ζητάει το λόγο και η κυρία Λίντα Μακάβαν. Ο Χόρτ Σνέλχαρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και θέλω να ξανανοίξω ένα θέμα που είναι η ενημέρωση της κοινή γνώμης. Πολλά ακούστηκαν και η παλέτα ε, είναι μια βεντάλια ολόκληρη το φάσμα αυτό από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσείς που εκπροσωπείτε τους καταναλωτές, ποιοι είναι οι καταναλωτές. Ιδρύματα, φορείς, σύνδεσμοι, πράγματα που χρηματοδοτούνται από διάφορες επιχειρήσεις για να βάλουν τρικλοποδιές στο δίπλανο. Και να διατρανώνουν διάφορα πράγματα και να εξαγγέλουν που δεν συμβαίνουν επίσημα. Ε, είπατε κι εσείς, ε, κύριε Μπιλόνι, να ε, κάνουμε μια διάκριση στον ορισμό της απάτης και της μη συμμόρφωσης. Εντάξει, η απάτη τότε να δημοσιοποιείται και η μη συμμόρφωση όχι, αυτό με προβληματίζει εμένα. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι ύποπτοι απάτης, όλες οι επιχειρήσεις από χέρι και εξορισμού. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο να δημοσιεύονται αυτόματα όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων γιατί μπορεί να απειληθεί και η επιβίωση της εταιρεία. Το σύνορο όμως αχωριστική γραμμή που είναι. Από ποια στιγμή δικαιούται μια κρατική αρχή, ένας επιθεωρητής να ε, δημοσιεύει. Γιατί κάθε δημοσίευση θεωρείται από την εταιρεία απειλή. Κρίμα που έφυγε εκπρόσωπο των καταναλωτών, γιατί είπε το σύστημα της διαπόμπευσης στη ε, Δανία της δηλήτευσης οδήγησε σε λιγότερες δηλητηριάσεις. Ε, στη Γερμανία δεν έχουμε το σύστημα αυτό, αλλά δεν έχουμε και δηλητηριάσει. Mm. Πώς το λένε αυτό, shame και κάτι, name ναι, and shame, εν πάση περιπτώσει. Κατονομάζεται ο και εκτίθεται θα ήθελα να έχω τη δική σας άποψη. Πώς το απαντάτε. Ε, τι θεωρεί η εταιρεία σας. Εντάξει, καλό αυτό που λέτε διάκριση, τι είναι απάτη και τι δεν είναι, τι είναι μη συμμόρφωση. Από ποια στιγμή και μετά όμως θα πρέπει να δημοσιεύεται το όνομα της εταιρείας. Και όταν ε, ε, έρχονται να σας ελέγξουν, εσείς θέλετε περισσότερες πληροφορίες από την εταιρεία ε, από την αρχή που σας ελέγχει για το πώς μπορείτε να βελτιωθείτε ή την έχετε ήδη αυτή την πληροφόρηση. Είναι απρόσκοπτη η συνεργασία σας. Και πού γίνεται ο έλεγχος, είναι ισορροπημένος. Ευχαριστώ. Η Λίντα Μακάβαν και μετά η κυρία Ράιμερ. Yeah, to... Uh, θα ήθελα να θέσω δύο ε, σημεία. Θα ήθελα η Επιτροπή να μας πει ε, ποια, ποιοι τομείς καλύπτονται από την οδηγία. Καλύπτουμε και τους ε, μεσάζοντες στον τομέα του κρέατος. Δεν νομίζω ότι καλύπτονται από την διατύπωση που υπάρχει όταν μιλάμε δηλαδή για οικονομικούς φορείς, για οικονομικούς φορείς τροφίμων. Μιλήσαμε λοιπόν και για τις επιθεωρήσεις που δεν προανακοινώνονται. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και η, η συχνότητα των ελέγχων, ιδιαίτερα στα, ε, στα διάφορες, διάφορες μονάδες κοπής κρέατος, όχι τόσο στα σφαγεία. Πώς έχει αυτό το θέμα της συχνότητας των ελέγχων. Ευχαριστώ κυρία Ράιμαρς. Ναι, μια που φτάσαμε ε, στους παραγωγούς τώρα, ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν σας έρχεται ο επίσημο έλεγχος, είτε είστε μεγάλη εταιρεία, επιχείρηση, είτε μικρή. Αυτό πώς επηρεάζει την εργασία, την καθημερινή και τι κόστος προκαλείται από τον έλεγχο. Αυτό δεν ακούστηκε ακόμα. Τη μέρα που έρχεται ο έλεγχος. Εγώ είμαι αγρότησα και ξέρω ότι ε, κάθε μέρα θα πρέπει να έχω στο μυαλό μου και να εφαρμόζω την ομοθεσία. Και όταν έρχεται ο έλεγχος στην ε, εκτροφή έρχεται να με ελέγξει για ένα νόμο, για ένα συγκεκριμένο. Και έτσι πολλαπλασιάζονται και οι έλεγχοι. Και όταν μιλάμε για αποτελεσματικού ελέγχου, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα και αυτό. Δηλαδή, σου έρχεται ο έλεγχο, αλλά σου δημιουργεί, σου προκαλεί και κόστο τη μέρα που έρχεται ο επίσημο έλεγχο. Γιατί είναι επιβάρηση αυτό για την εκτροφή σου. Και αυτό καλό θα ήταν να υποθεί καμιά φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Ε, θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση για να συμπεριλάβετε τις απαντήσεις σας. Ε, τώρα, όλο το απόγευμα κάπως συγκρουόμεθα για τη χρηματοδότηση, έτσι δεν είναι, των ελέγχων. Και προηγουμένω ακούστηκε μόλις, δεν θυμάμαι ποιο το είπε, κύριος Μπορέλο, ότι θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση στους ελέγχους που έχουν οικονομικές επιπτώσεις και ελέγχους που έχουν άλλες επιπτώσεις. Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ, με βασάνισε. Ποιος έλεγχος έχει και οικονομική ε, επιτυχία σε ό,τι αφορά ε, τις εταιρείες ή τις επιχειρήσεις κοπής κρέατος. Ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα το θετικό του κύριου ελέγχου. Και μετά ο κύριος Μπινόνι πήρε το λόγο και μίλησε για τον έλεγχο των σπόρων και τότε το κατάλαβα. Α, αυτός είναι ο έλεγχος που σημαίνει οικονομική επιτυχία, διότι εσείς λέτε ότι έχετε πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό και είστε ε, σε ηγετική θέση. Ε, είπατε ε, ότι θέλετε να έχετε και αυτό έλεγχο και αυτοπιστοποίηση και πάλι με προβλημάτισε αυτό. Τι σημαίνει. Αλλά σιγά σιγά άρχισα να το καταλαβαίνω και πήρα και την απάντηση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Όταν έχω μια εταιρεία και παράγω πιστοποιημένο σπόρο και κυκλοφορεί στην αγορά, τότε ο έλεγχος είναι εγγύηση για την επιτυχία μου και για τη θέση που έχω στην αγορά. Γιατί εάν είναι άχρηστος ο σπόρος, γιατί έχει μικρόβια, ιούς και δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπορώ να το πουλήσω μετά το σπόρο μου αυτό. Δηλαδή, έχει συμφέρον και ο παραγωγός και οικονομικό εννοώ συμφέρον να γίνονται οι έλεγχοι και οι αυτοέλεγχοι. Γι' αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το βλέπουμε και από αυτή τη σκοπιά και από τη διαφοροποίηση αυτή. Και πολλές μικρές επιχειρήσεις στη Γεωργία πραγματικά ε, επιβαρύνονται πάρα πολύ από τους μεμονωμένους ελέγχους. Το είπε τώρα και η Μπρίτα Ράιμερς. Και διερωτώ με. Γιατί είχα διατελέσει και συγκήτρια εγώ ε, για την προστασία του πολλαπλασιαστικού υλικού και την αηφόρο χρήση των σπόρων. Πάντα ζητούν ε, πιστοποιήσεις και αποδείξεις αηφορίας και ε, έλεγχη στην εκτροφή, για την διασταυρωμένη συμμόρφωση και όλα αυτά τα πράγματα συντονισμός δεν γίνεται να υπάρχει. Η κυρία Ράιμερς λέει ότι κάθε μέρα σου έρχεται ένας ελεγκτής για έναν άλλο νόμο. Και στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας συντονισμός όταν γίνεται έλεγχος να γίνεται. Άπαξ, δεν χρειάζεται να ξαναρθεί άλλος για άλλη νομοθεσία. Αυτά είναι τα ερωτήματα για την καλύτερη δυνατότητα συντονισμού ε, όλων αυτών των θεμάτων. Ο Σνάιχαρτ θέλει κάτι να προσθέσει και μετά απαντήσεις. Ναι, πρέπει πραγματικά να κάνω τη ε, σαφή, ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέμε ότι το πρόβλημα είναι τα οικονομικά. Ποιο είναι το ύψος του τέλους ε, που επιβάλλεται. Πώς κοστολογείται αυτό ε, όταν ελέγχει μια κρατική αρχή σου λέει έχω ένα κοστολόγιο 1000 ευρώ. Πώς το μοιράζω αυτό το χιλιάρικο. Όταν σε μια άλλη επιχείρηση κοστίζει αυτό 500 ευρώ. Πώς υπολογίζετε πώς το κοστολογείτε, είναι γενικά αναχώρα, αναπεριφέρεια, ανα εταιρεία. Εντάξει, μετά γίνεται ο οικονομικό έλεγχο. Αλλά πώς, πρώτον πώ υπολογίζεται το κόστο και μετά πώ επιμερίζεται το κόστο αυτό για του ελέγχου. Έχω ένα μικρό πρόβλημα εγώ σε αυτό. Ναι. Κύριε Ποντουλέ, σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα απαντήσετε αμέσω. Ε, πρώτα θα απαντήσουν οι κύριοι του τελευταίου πάνελ με τη σειρά. Πρώτο ο κύριο Καλντερόνε, παρακαλώ. Ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα για το πρώτο ερώτημα, για τη διαφορά μεταξύ απάτης και μη συμμόρφωσης. Πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι υπάρχει ένα σύστημα που υπάρχει, που υπάρχει και λέγεται σύστημα έγκυρης προειδοποίησης και που προειδοποιεί όντως τους ενδιαφερόμενους, τους, α, τις αρχές ελέγχου και του, τους επιχειρηματίες για τον ενδεχόμενο κίνδυνο για που προκύπτει όταν βάλει κανείς στην αγορά ε, κάποια τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα, που δεν είναι ασφαλή, υγιεινά κτλ. Με αυτόν τον τρόπο ε, εντοπίζουμε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αθέλητης, ε, αλλά και απάτης. Χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα σε ό,τι αφορά τη διατροφική ασφάλεια, ε, κίνδυνοι που από την κατανάλωση τροφίμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θέματα που δεν αφορά την ασφάλεια τροφίμων. Ε, Παραδείγματο χάρη, μιλήσατε τόσο πολύ για το πρόσφατο σκάνδαλο με το λογιστικό κρέα. Είναι μια απάτη κανονική, έτσι. Ε, δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων, έτσι. Δεν είναι ένα υγειονομικό θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα εμπορικό, έτσι. Πολύ σημαντικό. Ε, και δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου τη σημασία του θέματο αυτού. Στο δομέα του κρέατο ε, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έλεγχο. κατά τη σφαγή υπάρχει μόνη παρουσία του κτηνιάτρου. Τα κρέατα δεν μπορούν να τεθούν στο εμπόριο αν δεν έχουν την υγειονομική σφραγίδα, όπως λέμε. Είναι μια εγγύηση ότι έχει υπάρξει επίσημος έλεγχος. Στις επόμενες φάσεις παραγωγής, η μεταπητική βιομηχανία ε, που φτιάχνει προϊόντα με βάση το κρέας ε, και εκεί γίνεται έλεγχος σε εκείνο το επίπεδο και εκεί οι επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καταχωρημένες και να ελέγχονται. Δεν μπορεί δηλαδή μία επιχείρηση η οποία δεν ελέγχεται επίσημα κτλ. Ε, δεν μπορεί να βάλει στην αγορά τέτοια προϊόντα. Ε, για μας η διαφάνεια των ελέγχων δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Το εφαρμόζουμε ήδη. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για τους ελέγχους. Ε, αφού υπάρχουν τόσοι έλεγχοι, ας είναι και αποτελεσματικοί, έτσι δεν είναι. Κάτι που ξέχασα στην πρώτη παρουσίασή μου είναι να αναφερθώ στο θέμα τη εξαίρεση των μικρο... μικροεπιχειρήσεων, όπως προβλέπει η πρόταση κανονισμού. Ε, Εμεί ε... μεταξύ των μελών μα έχουμε και μικρέ τέτοιε επιχειρήσει. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Αυτέ οι εξαιρεσει δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στου εμπορευόμενου να έχουν του ίδιου ελέγχου, αλλά να μην συμμετέχουν στα έξοδα καθόλου. Να ελέγχονται δηλαδή χωρί να πληρώνουν. Όπως είπε σωστά και ο κ. Μπορέλο πριν, ε, επειδή έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις, τελικά τους ελέγχου τους πλέον αυτές οι πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε, στην, οι μεσαίες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ιταλία και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Ε, και τώρα περνάω στη τελευταία παρέμβαση. Εμείς έχουμε μια προϋπόθεση στην περίπτωσή μας όπως είπα για τους ε, ελέγχους, ε, για μας οι έλεγχοι στα κράτη είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, είναι μπανάλ γεγονός. Είναι υποχρεωτική και είναι ειδικά υποχρεωτική για τις εξαγωγές τρίτες χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ε, δεν λειτουργούμε χωρίς ελέγχους. εγώ θα μιλήσω Ιταλικά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία στο κόστος ελέγχων και την αξία τους για το τομέα των σπόρων. Ως προς τις δαπάνες στον τομέα των σπόρων θα ήθελα να πω ότι είναι αναλογικές οι δαπάνες ανάλογα με τον όγκο παραγόμενων σπόρων. Πρόκειται για συγκεκριμένο κόστος. Σας μίλησα για την αλυσίδα των ελέγχων που γίνεται στον τομέα αυτό και ε, το κόστος καλύπτεται ανατόνο ή κιλό. Άρα εμείς θεωρούμε ότι οι ΜΜΕ δεν κατακλείζονται ιδιαίτερα από αυτή τη φορολόγηση και υπάρχει μια δίκαιη κατανομή ε, κόστου στις ΜΜΕ. Υπάρχει λοιπόν μία ισοκατανομή ε, ως προς ελέγχου στον τομέα των σπόρων. Σε σχέση τώρα με την αξία των σπόρων που ελέγχονται, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να χρησιμοποιηθούν. Δεν υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα ως προς τους ελέγχους και το τελικό προϊόν, δηλαδή τον καταναλωτή που μπορεί να ενημερωθεί και να μπορέσει να αξιολογήσει τους σπόρους που έχουν ελεγχθεί. Άρα, ε, σε σχέση με το τομέα των σπόρων και τον τελικό καταναλωτή, θα μπορούσα να πω ότι οι σπόροι που ελέγχονται δεν αφορούν συγκεκριμένο προϊόν που φτάνει στο, στο πιάτο του καταναλωτή, αλλά υπάρχει ένα θέμα υγείας και υγιεινής που δεν καλύπτεται. Θα θέλαμε ως ιδιώτες να το προωθήσουμε και να υπάρχουν κανόνες έτσι ώστε να διοδίδονται οι πληροφορίες ως προς ελέγχους ε, στους οποίους υπόκεινται οι σπόροι για να δούμε ποιο είναι το εμπλεκόμενο κόστος το οποίο αφορά ε, το κόστος, το συνολικό κόστος που αφορά ολόκληρο τον, ε, τον τομέα μόνο, και να αφορά όχι μόνο τον αγρότη αλλά και τον καταναλωτή. Θα ήθελα να απαντήσω και σε αυτά που είπε ο προγενέστερος ομιλητής, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε τον καταναλωτή για να ξέρει τι αγοράζει. Αλλά ποιος θα ενημερώσει τους αγρότες. Μιλάμε για πολλές πληροφορίες και νομοθεσία και όλοι μιλάμε για αποστολή ελέγχων στην εκμετάλλευση, στην αγροτική εκμετάλλευση, αλλά κανένας δεν λέει πώς αυτή η, αυτές οι πληροφορίες, αυτή η πληροφόρηση μπορεί να μετατραπεί σε, ένα νέο, σε μια νέα νομοθεσία που να είναι χρήσιμη και για τον αγρότη. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Κλάς στη δική της παρέμβαση, Νομίζω ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει η συνέργεια δημόσιο-ιδιωτικού τομέα η βιώσιμη χρήση και η εφαρμογή στην αγροτική εκμετάλλευση και φτάνουμε και στην ασφάλεια τροφίμων. Τελικά. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι πώς θα προστατεύσω την αγροτική εκμετάλλευση έτσι ώστε ε, αυτά, αυτά τα φυτά ή σπόροι να οδηγήσουν σε, σε ένα ασφαλές τρόφιμο. Αυτό αφορά η ασφάλεια τροφίμων και η συνέργεια ε, δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Κύριε Κλάς, ε, μιλήσατε για την επιθεώρηση και κατά πόσο ε, μπορεί να λέξει τα πάντα, μα πώς να σας απαντήσω με μια ερώτηση. Πώς μπορεί ένας αγρότης να εφαρμόσει τα πάντα. Εάν μπορεί να το κάνει, τότε αυτό μπορεί να το κάνει και ένα σωστά καταρτισμένος επιθεωρητής. Η κυρία Ράιμερ μίλησε για το, το έμεσο κόστος. Δεν θα ήθελα να απαντήσω με αριθμητικά στοιχεία, αλλά με μια συλλογιστική γενικότερα. Εξαρτάται από τον έλεγχο. Εάν ε, θέλετε παραστατικά, έλεγχο παραστατικών, απλώς, μπορείτε να το κάνετε εκτός από την περίοδο θερισμού. Ως προς, το, τον, ως προς τις ε, διαδικασίες αυτές, αν δεν δουλεύουν οι μηχανές ε, κατά τη διάρκεια του θερισμού, δεν μπορεί να γίνει και ο έλεγχος. Στις εκμεταλλεύσεις μου απασχολούν περίπου 2.000 αυτό που έχει σημασία είναι να γίνονται παράλληλοι οι έλεγχοι. Αν φτάσουμε στην περίοδο συγκομιδής και ζητήσουμε έλεγχο παραστατικών, ο καλλιεργητής θα έρθει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει πρόβλημα με τον έλεγχο καθε αυτό, αλλά με τον χρονισμό του ελέγχου. Είτε είναι ε, προανακοινωμένος είτε όχι προγραμματισμένος είτε όχι. Θα πρέπει λοιπόν να συμπάσχουμε και με τους ε, καλλιεργητές σε αυτήν την περίπτωση. Ως προς το, τη στιγμή του έτους όταν τελειώσει η περίοδος καλλιέργειας ή σποράς και πριν από τη συγκομιδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ο έλεγχος. Όμως υπάρχει και η δεύτερη επιλογή, όπου υπάρχει ο έλεγχος του ελεγκτή, του επιθεωρητή. Και αν θέλουμε να είμαστε ε, σωστοί και νομίζω ότι η Κομισιόν ε, γνωρίζει το βελγικό σύστημα, αν θέλουμε να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί, λάβετε υπόψη τον έλεγχο των επιθεωρητών. Και εδώ σταματώ. Ευχαριστώ πολύ. Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς υπολογίζεται και πώς επιμερίζεται το κόστος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριο Σπούτλε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απαντήσω στην κυρία Μακάβαν. Μετά την κρίση του αλογίσιου κρέατος, διευκρινίσαμε τη νομική κατάσταση που ισχύει απέναντι στα κράτη-μέλη για τους εμπόρους, λεγόμενους traders ε, στο κρέας αλόγου. Υπήρχαν πάρα πολλοί ε, ενεχόμενοι traders. Αυτοί δουλεύουν, είναι δύο ειδών, είτε από το σπίτι τους με υπολογιστές που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε να τους επισκεφθούμε και υπάρχουν και κάποιοι traders που δουλεύουν με αποθήκες, ψυγεία και εκεί είναι πιο εύκολο. Παρόλο που οι εθνικοί επιθεωρητές ανέκαθεν θεωρούσαν τα ψυγεία και τις αποθήκες εκεί ως ένα τόπο που δεν γίνονται και πολλά πράγματα εάν γίνεται σεβαστή η θερμοκρασία. Ε, αν είναι στους μείον 18 βαθμούς συνέχεια, μέρα, νύχτα και όλο το χρόνο ε, και εκεί ο έλεγχος γίνεται μια φορά το χρόνο, θεωρούν οι ελεγκτές ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Δυστυχώς εδώ διαπιστώσαμε ότι στα ψυγεία τα ίδια, πράγμα που απαγορεύεται, αποσυσκεύαζαν τα κρέατα, έβαζαν, άλλαζαν τις ετικέτες, έκαναν ξανά τη συσκευασία και αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, οι trader αν έχουν ε, κατάψυξης και αποθήκες θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι, αν έχουν μόνο ε, υπολογιστή στο σπίτι τους θα πρέπει να είναι κάπου πιστοποιημένοι, δηλωμένοι. Αλλά θα πρέπει να έχουμε προσωπικό για να τους επισκέπτεται. Όταν είσαι trader και έχεις έναν υπολογιστή είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ο έλεγχος να σε βρει. Για το κόστος τώρα πώς ε, υπολογίζεται, ρώτησε ο κύριος Σνέλχαρτ. Η αρμόδια αρχή, κρατική είτε περιφερειακή, γιατί η Γερμανία έχει μια ιδιάζουσα κατάσταση, όπως και η Ιταλία και η Ισπανία που είναι χώρες όμως πονδού χαρακτήρα, θα πρέπει το κράτος να υπολογίζει το σύνολο του κόστους ε, των επίσημων ελέγχων αυτοκίνητα, εγκαταστάσεις, κατάρτιση, εργαστήρια και πάει λέγοντας. Και στη συνέχεια αυτό το κόστος θα πρέπει να ε, μετακυλίεται και με βάση το χρόνο ε, που ε, είναι κανείς σε μια επιχείρηση. Όταν έχεις ένα τυροπιτάδικο που χρειάζεται μισή ώρα ελέγχου, δεν θα πληρώνεις τα ίδια όταν είσαι, να είσαι μια επιχείρηση 250 ατόμων που παράγει κοιμά. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος, το ρίσκο εκεί είναι μεγαλύτερο. Λοιπόν, έτσι επιμερίζεται το κόστος, γίνεται ένας συμψηφισμός ανάλογα με το χρόνο που παραμένει κανείς στην επιχείρηση, ε, αλλά καταλαμβάνει και, και περιλαμβάνει όλο το κόστος, δηλαδή συμπεριλαμβάνει το μισό των επιθεωρητών. Αλλά οι επιθεωρητές δεν παίρνουν τα ίδια λεφτά στο βορρά της Ευρώπης και στο νότο. Για το λόγο αυτό λοιπόν δεν θελήσαμε να προτείνουμε ενιαίο τέλος ε, με ξέρω εγώ 50 ευρώ την ώρα για όλη την Ευρώπη. Αυτό μας είπαν αφήστε να το κάνουμε εμείς. Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, προσαρμογή στις τοπικές, περιφερειακές μέχρι και εθνικές συνθήκες. Εντάξει, αυτό το αφήνουμε στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη και να συνυπολογίζονται όλες οι παράμετροι. Και στο σύστημα που είχαμε για τις εξαιρέσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, δεν ε, τίθεται το θέμα να πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις τις μικρές. Τις μικρές επιχειρήσεις θα τις πληρώνει το κράτος σε καμία περίπτωση. Επειδή 90% των επιχειρήσεων είναι μικρές και δεν ελέγχονται, δεν θα πρέπει μεγάλες να τις πληρώνουν, σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός, ο περιφερειακός, ο τοπικός, ο δημοτικός, ο αρμόδιος. Επίσης θα πρέπει να γίνεται σεβαστή πάντα η ρύθμιση για τις κρατικές ενισχύσεις. Δεν θα πρέπει να γίνονται χάρες και ευνοϊκές μεταχειρήσεις στις πολύ μικρές επιχειρήσεις όταν πληρώνει το κράτος, η περιφέρει ο Δήμος. Στη συνέχεια, αυτό που ρωτήσατε εσείς κυρία Πρόεδρε, για το συντονισμό των ελέγχων των επιτοπίων στις εκμεταλλεύσεις. Αναφέρθηκαν και άλλοι σε αυτά. Και ο κύριος Πέτερς. Ναι. Η πρότασή μας τι στόχο έχει. Να είναι πιο συντονισμένες οι εθνικές αρχές όταν στέλνουν διάφορους ελεγκτές και επιθεωρητές επιφορτισμένους με διάφορα θέματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φυσικά είναι ανόητο να θεωρεί κανείς ότι θα έχει κάθε εβδομάδα καινούριο έλεγχο με ένα νέο ελεγχτή για να ελέγξει ένα ειδικό στοιχείο, ε, μια ειδική πτυχή της δραστηριότητας της γεωργικής της ε, κάθε εκμετάλλευσης. Αφήστε που δεν γίνεται και έτσι, αλλά εμείς τι θέλουμε, οι εθνικές αρχές να συντονίζονται και είναι ένας από τους στόχους του νέου κανονισμού. Πολύ καλύτερο συντονισμός έτσι ώστε ε, στις ε, εκμεταλλεύσεις όπως είπε ο κύριος Πέτερς να είναι ένας ο ετήσιος έλεγχος. Πρέπει να σας πω ότι οι αγρότες ήδη υφίστανται πολλούς ελέγχους. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό ο νέος ε, κανονισμός για τους αγρότες διότι ελέγχονται αυτοί ήδη για την πολλαπλή συμμόρφωση στην κοινή γεωργική πολιτική και πριν λάβουν τις επιδοτήσεις για να βεβαιωθούμε ότι υλοποιούν όλες τους κανόνες για την ευεξία των ζώων, για τον έλεγχο των ασθενειών, για τα φυτοφάρμακα κτλ. Γίνονται λοιπόν έλεγχοι και εστιασμένοι, ούτε πρόκειται να βελτιώσει τίποτα, αλλά κύριε Πέτερς, ναι, για τους γεωργούς και τους αγρότες το γνωρίζουν, θα πρέπει να μάθουν να σέβονται τους κανόνες, το είπατε, για τα φυτοφάρμακα και για την ευεξία των ζώων το κάνουν ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για αυτή την τελευταία σας απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση αυτή. Πολλά θέματα τα συζητήσαμε, πολλά ερωτήματα παρέμειναν αναπάντητα, προσθέθηκαν και άλλα ε, βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους συζητητές ε, Πυρίλο και Σνέρχαλτ που προείδρευσαν και στα δύο πάνελ του απογεύματος. Ευχαριστώ τους ομιλητές μας, άνδρες και γυναίκες και όλος ιδιαίτερος τον εκπρόσωπο της Λιθουανικής Προεδρίας ε, που παρέμεινε ε, και παρακολούθησε μέχρι τέλους το κύριο Κλουσίνσκας. Θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, δεν τελειώνει εδώ και ελπίζω κύριε Πυρίλιο να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Η έκθεση θα καταδεθεί αρχές Νοεμβρίου, τέλη Νοεμβρίου θα ξανασυζητηθεί εδώ στην Επιτροπή μας και μετά θα ψηφίσουμε το Γενάρη του 2014 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς. εμείς ευχαριστούμε. Κάνουν και υπερορίες, ε, όχι υπερορίες, υπερλεπτά, υπέρβαση ωραρίου, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ.